σας ενημερώνω ότι θα ότι η συνεδρίαση της Επιτροπής μας ε, μεταδίδεται απευθεία στο διαδίκτυο και στις γλώσσες που βλέπετε στην ενημέρωση που έχετε στα χέρια σας. Ερχόμαστε στο σημείο 3. Ανακοίνωση Επιτροπής, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεκτικό συνέδριο, συγγνώμη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο και Ελεκτικό Συνέδριο, περισσότερη λιγότερη έλεγχη, επίτευξη σωστή ισορροπία μεταξύ διοικητικού κόστου των ελέγχων και κινδύνου σφαλμάτων. Το λόγο έχει ο συγγητή μα ο κύριο Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε σε αυτή την. Αραιό ε, ε, κατοικημένη σήμερα Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Αλλά ξέρετε ότι οι σοσιαλιστές ε, λείπουν ε, για λόγους ε, εξωτερικής συνεδρίας που έχουν εκτός Βρυξελών σε μερίδες μελέτης. Θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι όμως που ενδιαφέρονται. Χαίρομαι που είναι εδώ ο κύριος Μετάρμοδης Επίτροπος και η κυρία Κάλλη Λάιτ από το Ελεκτικό Συνέδριο για να συζητήσουμε για το κίνδυνο των σφαλμάτων και τον ανοιχτό κίνδυνο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Σήμερα θέλω να σας πω ότι δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με το πώς, αλλά με το εάν μπορούμε καν να ε, συζητούμε για κίνδυνο σφάλματος και να ε, το αντιμετωπίζουμε. Γιατί δεν υπάρχει καν επιστημονικός ορισμός για το τι εστί κίνδυνο σφάλματος. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για τη γραφεία, τα έγγραφα συγγνώμη, εργασίας που μας έχει διανύμει στις διάφορες γλώσσες εργασίας. Έχουμε μια υπόθεση εργασίας, μια εισαγωγή και μια προϊστορία για το ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Επίσης ε, αναφέρεται εδώ στο έγγραφο το τι έχει κάνει μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο για τον ανεκτό κίνδυνο σφάλματος και επανέρχονται ε, και τα πολιτικά ε, ζητήματα, τα υπέρ και τα κατά σε ένα άλλο έγγραφο και προσπαθήσαμε να βρούμε εναλλακτική λύση στον ανεκτό κίνδυνο. Τροποποιούμε παλαιότερη απόφαση του Κοινοβουλίου του 2003, αλλά θα αναφερθώ στη συνέχεια σε αυτό εκτενέστερα worden. εισάγεται ήδη από το 2004 από το ελεκτικό συνέδριο η έννοια αυτή και να σας πω περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι τόσο πολύ το ανεκτό σφάλμα ή η ανεκτή απάτη. Είναι σχεδόν φιλοσοφική η έννοια ε, του ανεκτού κινδύνου σφάλματος όπως σας είπα αλλά δεν υπάρχουν σαφείς ακριβείς ορισμοί επιστημονικοί και για μας είναι σημαντικό ένα τέτοιο είδος κινδύνου, ένα τέτοιο κατόφλι αν θέλετε, να εισαχθεί. Γι' αυτό λέω συζητάμε για το εάν, εφόσον υπάρχουν αποδείξεις ότι όλα τα υπόλοιπα μέτρα έχουν ληφθεί για να αποφεύγονται σφάλματα. Ακριβώς εκεί λοιπόν βρισκόμαστε σε ένα προβληματικό σημείο. Το προβληματικό αυτό σημείο ποιο είναι. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα του Ελεκτικού Συνεδρίου σε πολλά σημεία σαφώς αποδεικνύει ότι τα συστήματα ελέγχου και διοίκησης των κρατών μελών δεν λειτουργούν. Και αυτό είναι οριστικό. Στο κεφάλαιο 4, σημείο 23, ε, παραπέμπει στο γεγονός του ελεκτικού συνέδριου ότι 30% των πόρων ε, δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί ε, λόγω και ελληματικών συστημάτων ελέγχου. Γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει. Ε, είναι τα πανηρά αυτά τα συστήματα ελέγχου και περίπλοκα και ταυτόχρονα χρειάζεται με εκπαίδευση, εκπαίδευση κατάρτιση για να προσαρμόζονται ε, στα ευρωπαϊκά στάνταρ και πρότυπα. Τα περισσότερα λάθη γίνονται στα κράτη-μέλη. Και υπάρχουν κράτη όπου κανείς υποπτεύεται ότι γίνονται πολλά λάθη, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα. Έχουμε όμως και καλές ειδήσει και στην αξιολόγησή μας ε, της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου και στη δική μου έκθεση. Εκφράσαμε την ικανοποίησή μας ε, για τη συνοχή. Δηλαδή το περιθώριο σφάλματος έχει μειωθεί από 11% στο 3% στις χώρες συνοχής. Ε, ήταν ευτυχείς οι περιστάσεις που επέτρεψαν κάτι τέτοιο. Γιατί χώρες που δαπανούσαν πολλά χρήματα και δεν ήταν και πάρα πολύ σχολαστικές ε, στον έλεγχο, αυτή τη φορά δεν ε, συμμετείχαν σε αυτό το θέμα. Και ποια είναι η καλή είδηση. Δεν είναι τύχη αυτό, ούτε ε, ακριβώς τυχαίο. Ε, οι αρμόδιοι επίτροποι διέκοψαν τις πληρωμές το 2009, δηλαδή δεν εκταμιεύθηκαν τα κονδύλια. Έγιναν έλεγχοι τυχαίοι σε χώρες όπως είναι η Ισπανία, ιδιαίτερα η Ισπανία και στην Ιταλία και δεν μπόρεσαν να εκταμιευθούν τα κονδύλια. Αυτό είναι καλή είδηση. Ε, οι μηχανισμοί ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργούν στο εσωτερικό της και ταυτόχρονα προχωρούν και σε διακοπή των εκταμιεύσεων. Ωραία όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Και αυτό είναι θετικό παράδειγμα. Αλλά παραμένουν ακόμα πολλά αρνητικά παραδείγματα που δεν έχουν εξαλειφθεί. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι στο βαθμό που τα ελεκτικά συστήματα και οι διοικήσει των κρατών μελών χωλένουν στην αποτελεσματικότητα, γιατί αυτό μας προσάπτει το ελεκτικό συνέδριο, υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο ελιγμών για βελτίωση χωρίς να αυξηθεί ο ανεκτός κίνδυνος φάλματος. Γιατί αυτό ε, υποθέτουμε εμεί και υποπτευόμαστε. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ επίπονο το έργο αυτό ε, για να βελτιωθεί. Και θα το πω τώρα με κάποια αφέλεια, αλλά και μια διάθεση προκλητική. Ε, αν αυξηθεί το περιθώριο αυτό σφάλματος, που τελικά δεν μπορεί να έχει θετική αξιολόγηση. Εμείς το βλέπουμε διαφορετικά. Ε, αντίστροφα, δηλαδή θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τα κακό σκήμενα και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Ποιο είναι τα κακό σκήμενα, ότι εξακολουθούν οι Υπουργοί Οικονομικών να ε, κάνουν τη δουλειά τους και να βάλουν και την υπογραφή τους. Δεν πέφτουν οι υπογραφές ε, ε στις ε, ε, δηλώσεις αξιοπιστίας των εθνικών διοικήσεων. Και εμεί καλούμε τα κράτη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Σουηδίας και των κάτω χωρών. Και εξακολουθεί να αρνείται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υπογράψει την έκθεση της θετική. Τα γνωρίζετε αυτά κύριε Σεμετά. μετά. Και επίση, Πώ να το πω, ε, εκθέσεις πεπραγμένων, ετήσιες και δραστηριοτήτων και πάλι δεν υπογράφονται από τους επιτρόπους. Επιπλέον πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει έναν αυτοματισμό σε χώρες που παραβιάζουν κατ' επανάληψη ε, τους κανόνες. Ακούστηκε επανειλημμένα εδώ το θέμα της Ελλάδας και ε, ε, το ΕΑΣ, το κτηματολόγιο που χρειάστηκε 10 χρόνια, 10 χρόνια που είναι πολύ ε, καιρό για να σταματήσει τις πληρωμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, δεν επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Αυτό που θέλουμε και αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα είδος αυτοματισμού, επαναλαμβάνω, που να μην επιτρέπει τα κράτη-μέλη να ασκούν πίεση και πολιτική επιρροή στην πολιτική απόφαση να σταματήσουν οι πληρωμές. Δεν ξέρω αν αυτό τώρα διακοπεί η ε, αναστολή interrupt, suspend, δεν ξέρω πώς θα τα πείτε αυτά νομικά, πείτε το πώς θέλετε, αλλά να υπάρχει μια αυτόματη διαδικασία και θα ήταν κάτι καινούριο αυτό να σταματάνε οι πληρωμές. Ε, και κάτι άλλο που μας ε, προβλημάτισε και συζητήσαμε ήταν μέτρα για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα ε, και της δουλειάς σας και να μπορεί να αξιολογείτε καλύτερα η έκθεση αξιολόγησης που έτσι και αλλιώς θα σας απασχολήσει από το 2011 λόγω της συνθήκης Λισαβόνας και έχουμε την αίσθηση ότι και εκεί υπάρχουν δυνατότητες να ε, αξιολογούμε καλύτερα τη δουλειά μας και εσείς την ίδια σας τη δουλειά καλύτερα με πολιτικούς στόχους που θα έχουμε από, μαζί, ε, από κοινού συγγνώμη, ε, και μαζί ορίσει για να κριθείτε και να μετρηθείτε σε αυτούς. Τώρα, στην επιστροφή πληρωμών των κρατών θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι συμβαίνει εκεί. Και σας παραπέμπω εδώ στους ετήσιους λογαριασμούς. Είναι μια έκθεση που είχατε την καλοσύνη για πρώτη φορά να δημοσιεύσετε με αυτή τη μορφή που σας δείχνω και για πρώτη φορά έχουμε κάποια εικόνα για τα όσα έπραξαν ή παρέλειψαν να πράξουν τα κράτη-μέλη. Και αν κοιτάξετε αυτού του ετήσιους ε, λογαριασμούς θα διαπιστώσετε ότι η Ισπανία στην προγραμματική περίοδο 2000-2006 στη συνοχή Δηλαδή όλα τα ταμεία που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικά και τα περιφερειακά ζητήματα έχει δηλώσει ε, διορθώσεις 2,5 δισεκατομμύρια. δηλαδή αχρεωστήτως καταβληθέντα είναι αυτά, 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ αχρεωστήτως καταβληθέντα στην Ισπανία και υποχρεώθηκαν να το διορθώσουν και να το επιβεβαιώσουν και να το αναγνωρίσουν. Για να δούμε τώρα τι μπήκε στον κορβανά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ουσιαστικά. 57 εκατομμύρια από τα 2,5 δις. Αχρεωστήτως καταβληθέντα. Μόλις 57 εκατομμύρια επέστρεψε η Ισπανία. Ε, είναι αξιοσημείωτη αυτή η ε, διάσταση και διαφορά και χαίρομαι ε, που αρχίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κατονομάζει και κράτη-μέλη. Μέχρι τώρα δεν το είχαμε δει αυτό και είναι ένας πρώτος δρόμο για να θέσουμε πολύ συνειδητά το δάκτυλο επί τον τύπο των ήλων και να πούμε φτάνει πια. Και αυτό λέει και το Κοινοβούλιο. Γιατί είναι καταφανώς προβληματικά αυτά τα νούμερα και τα κράτη που έχουν αυτή τη στρεβλή συμπεριφορά. σε έφερα την Ελλάδα, την Ισπανία, θα μπορούσα να μιλήσω και για την Ιταλία, για το κοινωνικό ταμείο. 24 έργα, για παράδειγμα, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προβλήματα. Ναι, ναι, ναι. Και στη Γερμανία. Ναι. Λυπάμαι πολύ αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Γιάλα. Το πρόβλημα της Ισπανίας είναι τόσο καταφανές που είμαι υποχρεωμένο να το αναφέρω. Είναι χρήματα των φορολογουμένων. Και οι φορολογούμενοι μας ψηφίζουν και εμάς, ψηφίζουν και εσάς. Και εγώ δεν έχω τώρα καμία όραξη να ρίξω το πέπλο της διπλωματίας από πάνω. Σας δώσω και το βιβλιαράκι να το διαβάσετε. Ευχαρίστω. Ε, το έχουμε επιτάπητο. ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι καιρός να ασχοληθούμε με τα στοιχεία. Και αναφέρω και τη Γερμανία γιατί στην περιφερειακή πολιτική η Γερμανία δεν μπορεί να στήσει ένα σύστημα ελεγκτικό στην περιφερειακή πολιτική. Γιατί, γιατί είναι χώρα ομοσπονδιακή. Το ίδιο πρόβλημα έχει και η Ισπανία και, ε, θα, ε, ε, και επιτίθεμαι και στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών και το κάνω που αρνείται να βάλει την υπογραφή του στη δήλωση εξοπιστία γιατί είναι χώρα ομοσπονδιακή και δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη. Να τα λέμε το όνομά του αυτά τα πράγματα. Αλλιώ δεν θα προχωρήσουμε. Σταματώ εδώ και λέγω. Η δική μας εναλλακτική πρόταση στο παρόν έγγραφο εργασίας μπορείτε να το διαβάσετε ε, φτάνει μέχρι το 2003 και παραπέμπει στην έκθεση απαλλαγής ε, ε, να έχουμε ένα κατάλογο κρατών μελών και τομέων πολιτικής που για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν πολύ σαφείς εκτιμήσεις και των σφαλμάτων αναχώρα για να δούμε και ποια είναι η ποιότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, γιατί διαφέρει από χώρα σε χώρα. Για να έχουμε ένα σαφές ε, δείγμα, μια σαφή εικόνα. Οι αιτήσιοι λογαριασμοί είναι πολύ καλό και χαίρομαι γι' αυτό και για το ελεκτικό συνέδριο που θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Με βάση αυτή τη μήτρα τώρα, αυτό το Matrix, έχει την ε, δυνατότητα να ε, αξιολογεί πολύ καλύτερα την ακρίβεια και το αληθές όλων αυτών των στοιχείων. Επίσης μπορεί να κοιτάξει και να παρακολουθεί καλύτερα και το σφάλμα που έχει διαπιστωθεί αλλά και τις επιστροφές που πραγματικά καταβάλλονται γιατί αυτό είναι το θέμα. Οι απαιτήσει ε, φτάνουν μόλις, μόλις στο 10% ε, να υλοποιούνται κύριε μετά και αυτό είναι πολλά λεφτά καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα χαιρόμουν πολύ σήμερα να μπούμε σε ουσιαστική συζήτηση και χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία της εκπροσώπου ε, του ελεκτικού συνεδρίου της κυρίας Καϊολάιτου, που είναι και εμπειρογνώμων. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε αμέσω το λόγο στον εκπρόσωπο του ελεκτικού συνεδρίου, την κυρία Να Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη του Κοινοβουλίου, Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να συμβάλλω με κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν τις ορισμούς, εκτίμηση και εφαρμογή της έννοιας του ανεκτού κινδύνου. Καταρχάς, όσον αφορά τον ορισμό, όπως ήδη είπε ο εισηγητής, το ελεκτικό συνέδριο στην γνωμοδότησή του το 2004, όσον αφορά το ενίο μοντέλο ενέχου, εισήγαγε την έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος και χρειάστηκε ισορροπία μεταξύ του κόστου του ελέγχου και των ωφελών που απορρέουν από τον έλεγχο μέσω τη του κινδύνου του σφάλματο. Το Ελεκτικό Συνέδριο είπε ότι χρειάζεται να είναι ρεαλιστή κανεί και ορθολογιστή όσον αφορά τα αποτελέσματα των ελέγχων. Και είναι βασικό θέμα. Τα, τα συστήματα ελέγχου δεν μπορούν να έχουν στόχο το μηδενικό κίνδυνο, όχι γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ δαπανηρό, αλλά επειδή επίση δεν είναι πιθανό ε, να επιτευχθεί κάποτε. Οπότε δικούμαστε στο γεγονό ότι κάποιο ε, ποσοστό σφάλματο πάντα θα υπάρχει όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τα διάφορα προγράμματα δαπανών. Τώρα όσον αφορά του σκοπού το ελεκτικό συνέδριο τόνισε στη γνωμοδότησή του ένα του 2010 ότι η επίτευξη μια ε, σωστή αξιόπιστη ε, εικόνα όσον αφορά ε, τι δαπάνε των προγραμμάτων θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ καλά όσον αφορά την έλεγχο του ρυθμιστικού καθεστώτο και του συστήματο διαχείριση τη Ευρωπαϊκή Ενώσης όσον αφορά την δαπάνη των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εξετάσει ποιε είναι οι αδυναμίε των υπαρχόντων συστημάτων για να λύσει το κόστο και το όφελο και σε ποιου τομεί πρέπει να γίνουν κάποιε αλλαγέ όπου η ανάλυση συμπεραίνει ότι δεν είναι πρακτικό να πετύχει κανεί επίπεδο υψηλό συμμόρφωση με τα διάφορα προγράμματα όσα έχουν, διάφορε επιλογέ φαίνεται ότι είναι διαθέσιμε. Αυτέ συμπεριλαμβάνουν την απλούστευση των διαφόρων κανόνων, των μηχανισμών, σχεδιασμών των προγραμμάτων, στενότερο έλεγχο ή να μπορούμε να ανεχόμαστε μεγαλύτερο επίπεδο μη συμμόρφωση ή να λύγουν να σταματούν οι δραστηριότητε. Πέραν αυτού, το λεκτικό Συνέδριο ήδη ανέφερε στο έγγραφο προβληματισμού του που απεστάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Μάρτιο του 2009 και εκεί έλεγε ότι οδήποτε σύγκριση μεταξύ των εκτιμωμένων ωφελών και του κόστου των ελέγχων θα πρέπει να βασίζεται στην εύλογη πεποίθηση ότι εφαρμόζονται αποτελεσματικά και αποδοτικά τα ελεκτικά προγράμματα και αυτό δεν ισχύει τώρα. Στην ετήσια έκθεση του 2009 που παρουσίασε ο πρόεδρος Καδέρα του Ελεκτικού Συνεδρίου την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθούν τα συστήματα διαχείρισης που είναι μόνο μερικώς αποτελεσματικά. Τώρα, οι εκτιμήσει για να υπάρχει σωστή απόφαση σχετικά με το τι μπορεί να είναι ανεκτό σαν κίνδυνο σφάλματο, κάποιο χρειάζεται έναν υπολογισμό του κόστου ε, των ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένη και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των κρατών μελών. Θα πρέπει επίση να γνωρίζει κανεί τη λειτουργία, τη σχέση δηλαδή μεταξύ του κόστου των ελέγχων και των σφαλμάτων που θα διαπιστώνει κανεί όσον αφορά του διάφορου ε, ελέγχου για τι δαπάνε Εμπειρικά Ξέρουμε ότι περισσότεροι έλεγχοι σημαίνουν λιγότερα λάθη, αλλά δεν μπορούμε να αποδείξουμε ακριβώ ποια μορφή έχει η καμπύλη αυτού του αποτελέσματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέτο ε, παρουσίασε μια πρόταση σχετικά με το ανεκτό επίπεδο σφάλματο στο σχέδιο ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Οπότε αυτή η πρόταση θα υπεχρέωνε και δεν θα επέτρεπε απλώ τι νομοθετικέ αρχέ να αποφασίσουν στο επίπεδο του ανεκτού κινδύνου σφάλματο στην ενδεδειγμένη ομαδοποίηση στοιχείων του προπολογισμού. Τώρα, πώς η νομοθετική αρχή θα προσπαθήσει να πετύχει αυτό το στόχο, υποθέτουμε εξετάζοντας ε, τα παρελθόντα επίπεδα σφαλμάτων, αλλά τα αποτελέσματα ελέγχου του 2009 ώστε να μας έδωσαν ακριβώς το μήνυμα το οποίο χρειαζόμαστε σε αυτή τη φάση των συζητήσεων. Δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυστηρή εφαρμογή των κανόνων και με τα εργαλεία τα αποτρεπτικά που έχει στη διάθεσή τη, ναι εννοώ τι οικονομικέ διορθώσει, μπορεί να πετύχει καλύτερα αποτελέσματα από το ίδιο μοντέλο ελέγχων. σω να δούμε μια αύξηση τη αποδοτικότητα έτσι. Πέρσι φαντάζομαι ότι η συζήτηση θα αφορούσε το πώ μπορούμε να έχουμε επίπεδο ε, μεταξύ 5 και 7% το επίπεδο κινδύνου για τα ταμεία συνοχή. Πού είμαστε φέτο, η εφαρμογή τώρα. Αντίθετα με αυτά που ανέφερα όσον αφορά του ενδεχομένου σκοπού τη έννοια, του ανεκτού κινδύνου, ε, το ελεκτικό συνέδριο πρέπει να δηλώσει την γνωμοδότησή του όσον αφορά την πρόταση τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να χρησιμοποιεί τον εκτό επίπεδο κινδύνου αποκλειστικά σαν βάση για να αποφασίσει ποιο επίπεδο ε, μη τακτική χρήση των πόρων θεωρείται σαν κάτι ανεκτό εκ των υστέρων. Η πρόταση δεν απαιτεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνήσει άλλα στοιχεία που σχετίζονται με αυτή την έννοια. Ε, το ελεκτικό συνέδριο στην γνωμοδότησή του 1 του 2010 συστήνει σαφώς την εφαρμογή διαφόρων αρχών όταν γίνεται αναθεώρηση των προγραμμάτων ε, δαπανών για να δούμε κατά πόσο υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη ε, αξία αν είναι σαφή η στόχη και το όλο πρόγραμμα αλλαλιστικό και όσο πιο απλό γίνεται. Και τέλος κατά πόσο είναι πολύ σαφής ο καθορισμός του ποιο είναι υπεύθυνο. Ε, εφαρμογή αυτών των αρχών μαζί με το επίπεδο σφαλμάτων που υπάρχει στα διάφορα προγράμματα αγαπανών μπορεί να δώσει ποιοτικέ πληροφορίε στι νομοθετικέ αρχέ όταν θα κάνουν αναθεώρηση υφισταμένων ε, προγραμμάτων δαπανών ή αποφασίζουν νέα προγράμματα και όσον αφορά τομεακέ νομοθεσίε στα πλαίσια των συζητήσεων για το νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό θα κοιτάζ, ήταν προσέγγιση προ το μέλλον όσον αφορά την εφαρμογή τη έννοια του ανεκτού επίπεδου κινδύνου. Κάτι που ενδείκνεται τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νέα νομοθεσία και κάνει ανάλυση συνεπειών αυτή τη νομοθεσία. Και τέλο, να πω κάτι όσον αφορά του διάφορου ρόλου και διάφορε ευθύνε. Το ελεκτικό συνέδριο στην Ομοδότησή του όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημοσιονομικού κανονισμού παρατηρεί ότι η έννοια των ανοιχτού επίπεδου κινδύνου βασικά αφορά το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτοί πρέπει να συζητήσουν και να αποφασίσουν. Και θεωρεί ότι αν η νομοθετική αρχή, και αν το κάνει αυτό, θέλει να καθορίσει όρια για τον εκτό επίπεδο κινδύνου, θα ήταν καλύτερο να το κάνει αυτό μέσω υπείου, νομοθεσία, νομοθεσίας, μέσω κατευθυντήριων γραμμών προσανατολισμών παρά μέσω νομοθεσίας. Από την άλλη πλευρά, ορισμός του υλικού χαρακτήρα των στοιχείων είναι κάτι που αποφασίζει ο εξωτερικό ελεγκτό. Το ελεκτικό συνέδριο πρέπει να ορίσει κάποιο όριο σύμφωνα με διεθνεί προδιαγραφέ ελέγχων. Αυτέ οι προδιαγραφέ απαιτούν ο εξωτερικό ελεγχτή να χρησιμοποιήσει επαγγελματική κρίση όταν αποφασίζει το επίπεδο αυτό του υλικού χαρακτήρα των στοιχείων στον έλεγχο και να μην εξετάζει μόνο τα μοδοποιημένα σφάλματα αλλά και τα ποσοστά των σφαλμάτων για να γνωρίζει κατά πόσο η γνωμοδότηση οπορία από τον έλεγχο πρέπει να τροποποιηθεί ή όχι. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Δώσουμε το λόγο τώρα στον Επίτροπο Σεμέτα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα και τη δυνατότητα μου δίνετε να παρουσιάσω την άποψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την έννοια του ανοιχτού κινδύνου σφάλματο. Η σημερινή ποια κατάσταση ποια είναι και ποια είναι η μελλοντική πορεία. Η έννοια του ανοιχτού πιπέδου κινδύνου αποφασίστηκε από το ελεκτικό συνέδριο στην γνωμοδότηση που δόθηκε το 2004 όσον αφορά το ενίο πρότυπο μοντέλο ελέγχου. Και εκεί η, γνωμοδότηση έλεγε ότι σε διάφορου τομεί του προπολογισμού πρέπει να εφαρμόζονται διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, κυρίω λόγω του τρόπου διαχείριση τη φύση των δράσεων και τη διάδραση που έχουν με του τελικού δικαιούχου. Έκτοτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επανειλημμένω εξέφρασαν το ενδιαφέρον του και την υποστήριξη για την διερεύνηση, περαιτέρω διερεύνηση τη ενία αυτή βάσει της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατόπιν τίματό σα, οι πρώτε προτάσει για την ανάπτυξη πέδρου, την έρευνα, ενέργεια και μεταφορέ και τι σχετικέ πολιτικέ παρουσιάστηκε φέτο τον Μάιο μαζί με τη συμπερίληψη τη ενία TRE στο δημοσιονομικό κανονισμό. Στις αρχές του έτους το ελεκτικό συνέδριο επανέλαβε την ανάγκη που υπάρχει να σχεδιαστούν οι έλεγχοι που θα είναι αποτελεσματικοί όσον αφορά το κόστος βάσει του κινδύνου και αυτό αναφέρθηκε στην γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου 1 του 2010 που βρισκόμαστε σήμερα. Στη συζήτηση όσον αφορά το ανοιχτό επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να βασιστούμε στην καλύτερη κοινή συνεννόηση επί των ενιών. Γι' αυτό προτείνω να επιστρέψουμε στα βασικά στοιχεία πριν να αξιολογήσουμε τα θετικά στοιχεία τη λόγω Κατά την άποψή μου, αυτή η έννοια θα πρέπει να θεωρηθεί σε ένα νέο εργαλείο που θα βασίζεται στο συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου των προγραμμάτων, στο περιβάλλον κινδύνου για τα προγράμματα και θα πρέπει το κόστο των ελέγχων να είναι ανάλογο των ωφελών παπορέων, ενώ να υπάρχουν και εύλογε διαβεβαιώσει ότι ο κίνδυνο των μη εντοπιστέντων σφαλμάτων παραμένει σε ένα αποδεκτό ποσοστό. Αυτό αντικατοπτρίζει σαφώς την σωστή δημοσιονομική διαχείριση, δηλαδή την αρχή του άρθρου 27 του δημοσιονομικού κανονισμού που βασίζεται κυρίως στις αρχές της οικονομίας και εξοικονόμησης μάλλον και αποδοτικότητας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ο κίνδυνος είναι ένα σημαντικό θέμα σε όλα τα προγράμματά μας και είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παίρνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη της. Περίπου 1,8 εκατομμύρια πληρωμές καταβάλουμε κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο σε διάφορους τομεί πολιτικής Κάποιες από τις πληρωμές καταβάλλονται άμεσα στους δικαιούχους, παραδείγματος χάρη στον τομέα της έρευνας. Η τεράστια πλειοψηφία των πόρων όμως πηγαίνουν σε εταίρους που εφαρμόζουν τα μέτρα, κυρίως τα κράτη-μέλη, τις αρχές των κρατών μελών, που καταβάλλουν τις πληρωμές στους τελικούς ε, δικαιούχους. Ο κίνδυνο των σφαλμάτων σε αυτέ τι πληρωμέ διαφέρει σημαντικά μεταξύ διαφόρων τομέων πολιτική, ανάλογα με την περιπλοκότητα τη νομοθεσία, το είδο του τρόπου διαχείριση και άλλου παράγοντε, που αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνο των σφαλμάτων είναι υψηλότερο σε άλλου τομεί από ό,τι σε άλλου. Ε, πιο συγκεκριμένα, προγράμματα υποκοινή διαχείριση, όπου οι πληρωμέ γίνονται ενάντια αξιώσεων από του τελικού δικαιούχου, ε, θεωρούνται πιο επικίνδυνο τομέα ε, αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται περαιτέρω όσον αφορά του περίπλοκου, αν υπάρχουν περίπλοκοι κανόνε επιλεξιμότητα. Σημειώσαμε πρόοδο όσον αφορά τη βελτίωση των ελεκτικών μα συστημάτων και μειώνοντα το ποσοστό σφάλματο. Το, η δήλωση εξοπιστία του 2009 είναι η πρώτη που το γενικό επίπεδο σφαλμάτων για όλο τον προπολογισμό είναι 2 με 5% σε αυτό το φάσμα. Στο, στην πολιτική συνοχή, μόνο εκεί έχουμε, είμαστε πάνω το 5% το 2009 και αυτό αποτελεί σημαντική απόκληση μάλιστα επίδοση καλύτερη από ό,τι τη δήλωση εξοπιστίας 2008. Επενδύσαμε σε πιο αποτελεσματικού ελέγχου, γι' αυτό είχαμε το αποτέλεσμα αυτό και απλουστεύσαμε του κανόνε σε κάποιου ε, τομεί. Ε, πιο συγκεκριμένα, καταβάλαμε πάρα πολύ μεγάλε προσπάθειε να κάνουμε καλύτερου ελέγχου, βελτιώνοντα ε, τον έλεγχο των κρατών μελών όσον αφορά τι πολιτικέ συνοχή και έχουμε καλύτερου ελέγχου για το 2007 μέχρι 2013. Και αυτοί οι κανόνε λοιπόν έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Επιπλέον διακόπτουμε πληρωμέ και αναστέλουμε πληρωμέ όταν διαπιστώνονται κάποιε ελλείψει. Παραδείγματο χάρη στι πολιτικέ συνοχή 40 προγράμματα έχουν διακοπεί επισήμω ή έχουν ανασταλεί επισήμω, ε, έχουν ανασταλεί διάμεσε πληρωμέ συνολικό ποσό 1,75 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε 15 αποφάσεις για να σταματήσουν οι πληρωμές. Το 2010 αυτός ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε. Αυτά, αυτές είναι πάντα δύσκολες αποφάσεις και η πίεση που ασκείται επάνω μας είναι πολύ συχνά πολύ μεγάλη αλλά κάνει το καθήκον της Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω ότι οι προσπάθειές μας οδηγούν σε σημαντική μείωση του ποσοστού σφαλμάτων στην πολιτική συνοχή. Να σας δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα σχετικά με το τι κάνουμε όταν διαπιστώνουμε κάποια προβλήματα, κάποιες ελλείψεις. Το 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενετόπισε ατασταλίες στη διαχείριση πόρων ΦΑΡ από δύο βουλγαρικούς εφαρμοστικούς φορεί. Άμεσο διορθωτικό σχέδιο δράση συμφωνήθηκε με τι βουλγαρικέ αρχέ για να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίε όσον αφορά τα ελεγκτικά συστήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέστηλε τι πληρωμέ αναμένοντα την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων από τι εθνικέ αρχέ. Όμω, η έλλειψη επαρκού πρόοδου από τι βουλγαρικέ αρχέ οδήγησε στην απόφαση Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει τι εξουσίε διαχείριση που είχε δοθεί στου δύο αυτού φορεί τον Ιούλιο του 2008. Αυτό οδήγησε σε σημαντική οικονομική απώλεια για την Βουλγαρία. Η απόφαση αναστολή αυτών των πόρων, διακοπή των πόρων, έστειλε σαφέ μήνυμα προ τα κράτη-μέλη, τι υποψήφιε χώρε και ενδεχόμενε υποψήφιε χώρε σχετικά με τη σημασία που έχει η ορθή οικονομική διαχείριση. Τέλος, επίσης ενημερώνουμε κάθε χρόνο λεπτομερώς στην ετήσια έκθεση αστυνομικών υπηρεσιών του αρμοδίου για τα αποτελέσματα των ελέγχων και πώ θα καλύψουμε τι αδυναμίε συμπεριλαμβανομένη και Αναφορά λεπτομερού σχετικά με το, την πορεία των κατών μελών. Όπω είπα την πασμένη εβδομάδα εδώ και στην Ολομέλεια, συμμερίζομαι την άποψη του λεκτικού συνεδρίου ότι τα καλά αποτέλεσματα για το 2009 δεν σημαίνουν ότι το ποσοστό σφάλμα των, ε, που έχουμε εκεί θέλουμε και στο μέλλον. Εκεί θα μείνει έτσι στο μέλλον αν δεν καταβληθούν προσπάθειε από του αρμόδιους οικονομικού φορεί και τα κράτη-μέλη και τι διαχειριστικέ αρχέ των κρατών μελών δεν θα μείνει τα επίπεδα το σφάλμα. Σε πολλού τομεί αυξήσαμε και τον αριθμό των ελέγχων ε, με στόχο τον εντοπισμό και άλλων σφαλμάτων. Παραδείγματο χάρη στην ανάπτυξη πέθρου τα κράτη-μέλη έκαναν περίπου 300.000 επιτοπίους ελέγχους το 2008 για το οικονομικό έτος 2009 και αυτό αντιπροσωπεύει 8% του συνολικού αριθμού των δικαιούχων. Το κόστος αυτών των ελέγχων ήταν περίπου 985 εκατομμύρια ευρώ δηλαδή 7,27% των δαπανών φεογγά. Όμως, το επίπεδο σφαλμάτων είναι ψηλότερο από το επιθυμητό. Άρα δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τον αριθμό των ελέγχων και μόνο. Αυτό κοστίζει χρήματα και θέτει και άχθος επί των δικαιούχων για την έρευνα, την ενέργεια και τις μεταφορές η ανάλυση μας δείχνει ότι εν συγκρίση με το επίπεδο 3% των σφαλμάτων για να πετύχουμε το 2% που έχει τεθεί σαν στόχος θα μας κόστιζε άλλα 90 με 150 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για τους επιτόπιους ε, ελέγχους. Αυτή δεν είναι μια αποδοτική όσον αφορά το κόστος προσέγγιση και δεν κατοπτρίζει επαρκώς την αρχή της ορθής οικονομικής ε, διαχείρισης. Το θέμα πρέπει να εξετάσουμε μαζί σήμερα είναι κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να εξετάσουμε το δεχόμενο περαιτέρω απλούστευση και τα επόμενα προγράμματα σχεδιαστούν βάσει των αποτελεσμάτων αντί των ίσρων. Και θέλουμε ελέγχου που να βασίζονται στου κινδύνου, να είναι αποτελεσματικοί έλεγχοι στο κόστο και να παρέχουν τι διαβεβαιώσει ότι οι εγγενεί κίνδυνοι ε, μειώνονται επαρκώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένως ανέφερε ότι εδώ δεν μιλάμε για κατάσταση το επίπεδο υλικού χαρακτήρα των στοιχείων του εξωτερικού ελεγχτή που χρησιμοποιούν για τους ελέγχους τους. Θέλουμε να έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς εμείς που θα βασίζονται στην γνώση των δαπανών, των ωφελών και των συγκεκριμένων κινδύνων που δημιουργούνται σε τομείς προγραμμάτων. Η νέα στρατηγική των ελέγχων δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο ε, στην έμεση διαχείριση πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα προγράμματα διαχείριση, κυρίω στην κοινή διαχείριση, οι άλλοι οικονομικοί φορεί θα έπρεπε να δεσμεύονται από την υποχρέωση να εφαρμόζουν του ελεγκτικού μηχανισμού, ούτω ώστε να δίνουν επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι οι κίνδυνοι καλύπτονται επαρκώς με έναν τρόπο που είναι αποτελεσματικό όσον αφορά το κόστος. Αυτό που σχετίζεται και με την πρόταση που κάναμε όσον αφορά την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού να υποχρεώνονται οι εθνικές αρχές πληρωμών στα διαθετικά ταμεία κάθε χρόνο να εκδίδουν μια δήλωση αξιοπιστίας όσον αφορά τη διαχείριση που θα βασίζεται και σε μια γνωμοδότηση των ελεκτικών αρχών. Μας είπε το Συνέδριο ότι σε ανοιχτό επίπεδο επίπεδο κινδύνου και μια τέτοια προσέγγιση μπορεί να καθοριστεί η πυκνότητα των ελέγχων, συναρτήσει του κόστου και των ωφελών των ελέγχων και το επίπεδο των εκτού κινδύνου θα μπορούσε να ποικίλει μεταξύ διαφόρων τομέων του προπολογισμού, συναρτήσει των εγενών κινδύνων και του κόστου των ελέγχων. Αυτό θα εξασφαλίζει πραγματική μετακίνηση προ ελέγχου που είναι αποδοτική όσον αφορά το κόστο, παρά να προσπαθούμε να πετύχουμε ένα στόχο ιερό του 2% σε όλου του τομεί. Να μην λησμονούμε επίση ότι το κόστο των ελέγχων και οι ενεί κίνδυνοι όσον αφορά τα σφάλματα για τα προγράμματα δεν αποτελούσαν επίσημα τμήμα των συζητήσεων επί τη ε, παρούσα ε, νομοθεσία. Η δήλωση αξιοπιστία είναι αιτήσια, ενώ τα περισσότερα προγράμματα είναι πολιτή. Αυτό σημαίνει ότι κάποια σφάλματα βρίσκονται και διορθώνονται αφού κλείσουν αυτά τα προγράμματα και έτσι μπορούμε να μειώσουμε τα υπόλοιπα σφαλμάτων σε, μια, σε μεταγενέστερο στάδιο. Από ότι ε, διαπιστώνεται το επίπεδο σφαλμάτων στην ετήσιο έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου. Εξετάζεται ο κίνδυνο επιτήσια βάσεω και θεωρείται ω βάση όσον αφορά το επίπεδο του κινδύνου και μη εντοπιστέντων σφαλμάτων για το έτος αυτό το οποίο ελέγχεται. Οι έλεγχοι που γίνονται εκ των υστέρων θα επιτρέψουν διορθώσει των σφαλμάτων που δεν έχουν βρεθεί κατά το οικονομικό έτος, κατά το οποίο έκανε τον έλεγχο το ελεκτικό συνέδριο. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται επί της βάσεως ο ελεκτικός μηχανισμός. Στόχος. Το επίπεδο εναπομενών των σφαλμάτων στο τέλος των προγραμμάτων θέλουμε να παραμένει ε, χαμηλό. Πώς το TRE συνδυάζεται με, το, με την απλούστευση. Ένας το ελεκτικό συνέδριο ότι ε, είναι περίπλοκοι οι κανόνε επιλεξιμότητα και αυτό δίκη σε σφάλματα. Καθώ και οι κανόνε για τι δημόσιε προμήθειε στα ε, διαθετικά ταμεία και οι επενδυτικέ δαπάνε των δικαιούχων. Η απλούστευση των κανόνων επιλεξιμότητα θα μπορούσε να είχε επωφελεί συνέπειε όσον αφορά τα ποσοστά σφάλματο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επίση ότι η απλούστευση των κανόνων επιλεξιμότητα είναι σημαντικό παράγοντα για τη μείωση των κινδύνων σφαλμάτων σε μελλοντικέ πολιτικέ ε, σε διάφορου τομεί. Ταυτόχρονα σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι κανόνες είναι απαραίτητοι για να εξασφαλίζουν ότι οι συγκεκριμένοι στόχοι πολιτικών επιτυγχάνονται. Είναι σαφές ότι όλοι οι συμμετέχοντες φορείς θέλουν καταρχήν απλούστευση. Η πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής Ήτρε όσον αφορά την απλούστευση της εφαρμογής των προγραμμάτων πλαισίων για την έρευνα τονίζει και παραθέτω ότι η διαχείριση των ερευνητικών πόρων που διατίθεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και να ανέχονται κάποια επίπεδα κινδύνων ε, όσον αφορά συμμετέχονται σε διάφορα στάδια των προγραμμάτων και θα εξασφαλίζεται βέβαια και ο έλεγχο. Τέλο τη παράθεση. Χρειαζόμαστε να εξασφαλίσουμε ότι όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει συγκεκριμένε προτάσει, υπάρχει μια κοινή συνεννόηση όσον του στόχου τη πολιτική, του εγγενεί κινδύνου και ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να μειώσουμε το κόστο και τα επίπεδα των σφαλμάτων που δημιουργούνται από πολύ περίπλοκου κανόνε. Το να έχουμε μια βάση για συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα να, το Δεκέμβριο του 2010 θα υποβάλει ανακοίνωση η βάση των συζητήσεων και θα είναι και το πλαίσιο των συζητήσεων με τι νομοθετικέ αρχέ. Το ανεκτό επίπεδο σφαλμάτων δεν είναι κάτι αντιφατικό, ούτε αποκλείει την ε, απλούστευση αλλά είναι εξισορροπητικός παράγοντας μεταξύ περίπλοκου χαρακτήρα των διαφόρων νομοθετικών διατάξεων που ισχύουν σήμερα και από την άλλη ε, του κόστου των ελέγχων. Θεωρώ ότι μια προσέγγιση που βασίζεται σε κατανόηση των ελέγχων που βασίζονται στον κίνδυνο και που είναι αποδοτική όσον αφορά ε, το κόστος είναι σωστή βάση για την αξιολόγηση τη διαχείριση του κινδύνου πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλων οικονομικών φόρων. Λοιπόν, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφέστατη την άποψή τη και μα έχετε ενθαρρύνει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Και έτσι υποβάλαμε τι προτάσει που έχετε μπροστά σα. Για την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω πρέπει να αποφασίσουμε πώ θα λάβουμε υπόψη του κινδύνου που δημιουργούνται από την νομοθεσία σε αυτή την περίοδο και που θα έχει αποτελέσματα στην απαλλαγή που θα δοθεί μέχρι το 2018. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει τις βελτιώσεις της αποδοτικότητας ανέχου όπου αυτό είναι δυνατόν και θα εξακολουθεί να ασκεί πίεση από τον κρατών μελών να κάνουν το ίδιο. Θα καλύψουμε τις αδυναμίες κυρίως διακόπτοντας και αναστέοντας πληρωμές ε, και προβαίνοντας σε ανακτήσεις σπόρων χρειάζεται να είμαστε αυστηροί στον αφορά τα ελεκτικά συστήματα και πόσο ποτικά είναι όσον αφορά το κόστο. Θα συνεχίσουμε το διάλογο με τι νομοθετικέ αρχέ για να βρούμε μια λύση για να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα. Δηλαδή, σε κάποιου τομεί το κόστο τη επίτευξη του στοιχείου, του ορίου 2% είναι απαγορευτικό και δεν είναι συμβατό με την αρχή τη ορθή δημοσιονομική διαχείριση. Δεν θέλουμε επιταγή εν λευκό για θετική δήλωση αξιοπιστία ή να κάνουμε λιγότερου ελέγχου, χειρότερου ελέγχου. Ήδη δείξαμε ότι είμαστε αφοσιωμένοι στην προσπάθειά μα να βελτιώσουμε του ελέγχου Αυτό που χρειαζόμαστε είναι εύλογο όριο, λογικό όριο, για να μπορούμε να προσμετράμε βάσει αυτού τις επιδόσεις μα. Περιμένουμε από εσά τη συνέχιση του διαλόγου του θέματο αυτού και να βρείτε μια λύση για την περίοδο μετά την νομοθεσία που λήγει το 2013 και που θα επηρεάσει τι δηλώσει αξιοπιστία. Βασιζόμαστε στην υποστήριξή σα επίση να εισαγάγετε πιο ισχυρέ διατάξει όσον αφορά την διαχείρισης, τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό και να πετύχεται μέγιστη απλούστευση μετά το 2013, κάτι που θα έχει πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά τις δηλώσεις αξιοπιστίας και το επίπεδο των σφαλμάτων. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, Επίτροπο Σεμίτα. Ξεκινάμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους. Ο κύριος Ιτάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο Χατζημαρκάκη. Όντως εδώ τίθενται πολλά ερωτήματα, για τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε και μια απάντηση. Καταρχάς, αν όντως η προσθέμενη αξία των περισσότερων ελέγχων θα μπορέσει να φανεί και στους ε, ε, φορολογούμενους. Μετά, το ερώτημα των δικαιούχων των ε, πόρων. Αν μπορεί να, όντως να ε, υπάρξει η δυνατότητα υπολογισμού λιγότερων λαθών. Και μετά τι γίνεται με τις... Ε, ποιες είναι οι συνέπειες όταν αυξηθεί αυτός ο ανεκτός κίνδυνος φάλματος ή το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. Τι μήνυμα δίνει αυτό το ενδεχόμενο. Θέλουμε φυσικά να ε, βελτιωθεί η αξιολόγηση των σύνολό τη. Και μετά, πώς ακούγεται για τους ψηφοφόρους, για τους φορολογούμενους όταν λέμε ότι το, ο κίνδυνος ασφάλματος δεν είναι μηδενικός. Δεν θα πρέπει με οποιοδήποτε μέσο να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα μηδενικό ή όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν κίνδυνο σφάλματος. Γιατί ξέρουμε ότι ακόμη και τα μικρά λάθη ε, παρισφρίουν στα ΜΜΕ και λαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη ε, σημασία από όσοι έχουν. Και μετά ο κύριος Χατζημακάκης ε, είπε κάποια πράγματα για την πολιτική συνοχή για τις αξιολογήσεις που γίνονται εκεί. Θα πρέπει και εδώ να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν, όπως είπα, πολλά Ρωτήματα τα οποία ακόμη είναι εκρεμή και βεβαίω θα πρέπει να τα απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Γιάλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστώ τον κύριο Χατζημαρκάκη. Αν και όπως πάντα μίλησε για την Ισπανία και για απόλυτους αριθμούς, όχι για ποσοστό, γιατί είναι το 3% το ποσοστό αυτό. Και υπάρχουν και άλλες χώρες με αντίστοιχα ποσοστά ε, στην πολιτική συνοχή. Βεβαίως θα πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά και η Ισπανική κυβέρνηση πέρσι συνεργάστηκε και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο μας για να βελτιωθούν τα συστήματα εκ των προτέρων ελέγχου που ήταν κάπως προβληματικά. Νομίζω ότι φέτος λειτουργήσε καλά και εν πάση περιπτώσει το είπα. για να είμαστε σωστοί και ακριβείς, να μην μιλάμε για απόλυτους αριθμούς, αλλά για ε, ε, ποσοστά. Είναι 3%. Ενώ η Γερμανία στο παρελθόν είχε λιγότερα κονδύλια, αλλά περισσότερο και μεγαλύτερο επίπεδο σφάλματος. Να μην τα ξεχνάμε αυτά και να συγκρίνουμε πράγματα και μεγέθη συγκρίσιμα. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα και εγώ να πω ότι θέλουμε να είναι όσο γίνεται λιγότερο το σφάλμα και ε, ο κίνδυνος. Βλέπουμε και τα έγγραφα εργασίας του ε, εισηγητού και ε, εγώ το βλέπω ως ένα επιπλέον μέσον για την ε, αύξηση της διαφάνειας και της ορατότητας προς τους πολίτες. Αλλά δεν υπάρχει αυτός ο ιδεατός κόσμος του μηδενικού σφάλματος και του μηδενικού λάθους. Πρόκειται για λογιστικά συστήματα και όταν μετράς κάποια μεγέθη ε, είναι πολύ δύσκολο ακόμα και από πολιτική σκοπιά να εξηγήσει κανείς πώς λειτουργούν αυτά τα λογιστικά συστήματα. Ευχαριστώ πάντως το Ελεκτικό Συνέδριο που έκανε την προσπάθεια να μας ε, παρουσιάσει και τους κινδύνους και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες από το νέο αυτό ε, κείμενο. Το θέμα είναι όχι απλώς να μας διευκολύνει, αλλά να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να απλουστευτεί το σύστημα για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες περί τίνος πρόκειται. Γιατί δεν είναι ο ίδιος ο κίνδυνος, ας πούμε, στο κοσυφοπαίδιο ή ε, ε, αλλού κάποιες περιοχές που έχουμε πάει ε, που είναι πολύ εκτεθειμένες οι περιφέρειες και δεν μπορούσε κανείς να κάνει τους ελέγχους με τον ίδιο τρόπο όπως γίνονται στις άμεσες πληρωμές. Το ίδιο ισχύει και συμβαίνει και στις ε, χώρες ε, σαν τις δικές μας που είναι ομοσπονδιακές. Όχι να μην γίνονται έλεγχοι, έλεγχοι γίνονται και βελτιώνονται, αλλά τελικά αυτό που λείπει είναι η υπογραφή. Η γενική, τελική υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών. Όταν τα συστήματα και το πολιτικό και το αποκεντρωμένο σύστημα είναι τέτοιο ώστε, πώς να το πω, δυσκολεύει πάρα πολύ την τελική υπογραφή του Υπουργού. Δεν είναι τυχαίο ότι γίνεται λόγο για τη Σουηδία και την Ολλανδία, αλλά η Σουηδία και η Ολλανδία δεν συγκρίνονται ούτε με τη Γερμανία ούτε με την Ισπανία ω προ τη δομή του κράτου. Έτσι, να προχωρούμε με μεγέθη συγκρίση, με επαναλαμβάνω, και να γίνεται παντού ο έλεγχο και στην πολιτική διαχείριση και στι πιστώσει ε, πληρωμών, αλλά και στην ανάληψη υποχρεώσεων, αλλά να προτείνουμε πράγματα που να χρησιμεύουν και σε χώρε τύπου ομοσπονδιακού. Γιατί δεν μπορούν να βρουν εφαρμογή συστήματα τύπου Σουηδία και Ολλανδία σε τέτοιε χώρε. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο σημείο 9, στο τρίτο έγγραφο εργασίας, ο εισηγητής λέει ότι τα κράτη-μέλη Μάλλον λέει, οι εθνικέ κυβερνήσει δεν είναι δυνατόν να κληθούν να λογοδοτήσουν για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται του πόρου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί είναι αυτή η τοπάθεια, δεν κατάλαβα. θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή στον προβληματισμό και να θεωρούν ότι βεβαίω του αφορά αυτό και θα πρέπει ε, οι πολιτικοί ηθήνοντε να λογοδοτούν και για το ε, τρόπο με τον οποίο απορροφούν τα κονδύλια γιατί αυτό το έλλειμμα διονίζεται και το ρίχνει τον μπαλάκι ο ένας στο γήπεδο του άλλου και τελικά ούτε το Συμβούλιο δεν μπορεί να εγγυηθεί ε, τη σωστή λειτουργία. Ενισχυμένη λοιπόν συνεργασία, ενισχυμένο διάλογο πλέον μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων και το Ελεκτικό συνέδριο, το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Ελεκτικά Συνέδρια. Μέσα σε όλο αυτό το διάλογο λοιπόν και τον προβληματισμό που μα ανοίγει μεγάλε ευκαιρίε για να βρούμε ποια είναι τα καλύτερα συστήματα, να προχωρήσουμε. Όχι μόνο για το κόστο καλύτερα, έτσι, αλλά και ω προ την αποτελεσματικότητα καλύτερα. Να προλαμβάνονται οι. Ε, καταστάσεις αυτές και τα σφάλματα και να μην τρέχουμε να τα διορθώνουμε εκ των υστέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γκέιρ, ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σχολιάσω και εγώ κάποια πράγματα. Η Κομισιόν όντως ε, σωστά έπραξε με τον ανεκτό αυτοκίνδυνο σφάλματος ε, που θέλει να κοιτάξει για κάθε πρόγραμμα συγκεκριμένα ποιος είναι. Το έφερε και η κυρία Αγιάλα. Φυσικά είναι σαφές αυτό, γιατί ούτως ή άλλως θα μιλήσουμε και για τη διεθνή βοήθεια. Ο, εκεί ο ανεκτός κίνδυνος σφάλματος είναι διαφορετικός όταν μιλούμε για άμεση βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες, ε, από ότι ας πούμε στην ε, χρηματοδότηση της έρευνας οι αναπτυσσόμενε χώρε ε, ε, και αυτές έχουν πρόβλημα στην ε, δημόσια διοίκησή τους, οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα χειριστούν τα δημόσια οικονομικά τους όπω θα διαχειριζόμαστε εμεί, α πούμε, όπω θα το επιθυμούσαμε εμείς εδώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει όμω μπορούν έτσι σε πρώτο επίπεδο Τη ανάλυση να δούμε, μπορούμε να δούμε ποιος είναι τελικά αυτός ο ανεκτός κίνδυνος φάλματος. Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο σε μια τριμερή συζήτηση, να ξεκινήσουμε μια τριμερή συζήτηση με το Συμβούλιο. Γιατί, Γιατί και τους αφορά, ή θα έπρεπε να τους αφορά, να υπάρξει συμβόλαιο δηλαδή, για το πώς ε, Πώ μπορεί να μειωθεί ο ανεκτός κίνδυνο του Σφάλματο για την Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον. Δεύτερον, μπορούμε να καταδείξουμε νέα λάθη, αν δεν έχουν καταγραφεί. Εγώ ε, κάνω και την αυτοκριτική μου όταν βλέπω, α πούμε, στα δείγματα, στα δείγματα που κάνει το ελεκτικό συνέδριο, δεν υπάρχει κανένα ε, γερμανικό σύστημα ελέγχου, το οποίο να είναι πλήρως αποτελεσματικό. Στην καλύτερη, στην καλύτερη περίπτωση, εντάξει, είναι στα όρια και εγώ ως ε, Γερμανός και ως Ευρωβουλευτής ενδιαφέρομαι και στα γερμανικά κρατήδια να ξεκινήσει μια συζήτηση για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω. Να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να συμβάλλουμε για να βελτιωθεί η κατάσταση στο μέλλον. Να μπορέσουμε αυτό τον κίνδυνο ασφάλματος να τον μειώσουμε. Και γι' αυτό θα ήθελα και με βάση όλα αυτά να μιλήσουμε για το τι ακριβώς σημαίνει αυτός ο ανοιχτός κίνδυνος ε, ασφάλματος. Τι καταλαβαίνετε τελικά ε, εσείς και πώς μπορούμε τελικά να καταλήξουμε σε τέτοιες εκθέσεις οι οποίες θα έχουν την υπογραφή ε, των υπευθύνων στο τέλος. Κύριε Επίτροπε, ο τρόπος ε, της, που κινείται η Κομισιόν είναι λίγο ασθενικός θυμάμαι την ανακοίνωσή σας και την έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά και όντως ε, λέτε ότι το κόστος ε, του ελέγχου με τα μέσα που θα, μπορούσε να έχει, που θα μπορούσαν να υπάρχουν για την, και, να, και τα λάθη που θα μπορούσε να ελεγχθούν, ότι θα πρέπει να ε, είναι συγκρινόμενα τα μεγέθη αυτά. Εντάξει, ως εκεί καλά. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική πτυχή του ανεκτού κινδύνου σφάλματος. Και κυρίως επειδή δεν μιλάτε για ανεκτό κίνδυνο σφάλματος. Μιλάτε για έναν ανεκτό, ένα ανεκτό ποσοστό σφάλματος. Και αυτό είναι κάτι άλλο. Μέσα στα έγγραφά μας, το θέμα των αποτελεσματικών ελέγχων και των αποδοτικών ελέγχων είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό σημείο. Αλλά κατά την άποψή μου δεν νομίζω ότι είναι το μόνο. Το είπαμε και στην αρχή, το είπα, αλλά και για πολύ απλούς λόγους δεν μπορεί να είναι το μόνο. Μερικές φορές είναι σκόπιμο να, έτσι, να υπερβάλλουμε και να τονίζουμε τις αδυναμίες μας. Το κόστος ε, ενός ε, οικονομικού ελεγκτή προφανώς είναι σημαντικό όταν κάνει τις, ε, τους ελέγχους του αλλά μπορεί αυτό να αυξηθεί και κατά 100%. Το κόστος φυσικά των ελεγχών είναι σημαντικό, αλλά αυτό δεν μπορούμε να το εντάξουμε στο πλαίσιο του ανεκτού κινδύνου. Δεν μπορεί να εννοούμε αυτό δηλαδή. Και απ' την άλλη δεν πρόκειται φυσικά να επιτύχουμε τον α, ιδεατό κόσμο όπου ο κίνδυνος λάθος θα είναι μηδενικός. Προφανώς δεν μπορούμε να καταλήξουμε στα δύο άκρα και δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να το επιζητούμε. Αλλά νομίζω ότι εάν μιλούμε για έναν ανεκτό κίνδυνο σφάλματος κατά την άποψή μου, είναι το πιο δαπανηρό λάθος. Το πιο δαπανηρό σφάλμα που θα πρέπει να αποφευχθεί. Και όχι αυτό που συναντάμε καθημερινά ή που είναι το πλέον σύνηθες. Ή ένα, ένα ε, σφάλμα που μπορεί να προκύπτει από το ίδιο το σύστημα. Ο ορισμό λοιπόν αυτού του ανεκτού κινδύνου σφάλματο θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο και να μην μιλάμε μόνο για το κόστο των ελέγχων. Το ελεγκτικό συνέδριο είπε, ε, μίλησε για το πόσα ε, λάθη γίνονται, πόσα σφάλματα γίνονται στι δημόσιε προμήθειε. Και συχνά έχουμε ασχοληθεί με τον τομέα αυτό είναι μια ζούγκλα από, προ, διατάξεις που όλες έχουν έναν στόχο να μειωθεί, να αποφευθεί η χειραγώγηση. Όλα καλά ως εδώ. Αλλά στον τομέα αυτό, ας πούμε, της Βόρειας Ιρλανδίας βασφαλίας αν κάποιος ε, δεν, ε, έχει, αν, κάτι δεν γίνει σωστά, τότε θα έχει, θα γίνει ένα λάθος. Μπορεί αυτό να θεωρηθεί ε, ανεκτό, λάθος γιατί δεν προκαλεί ε, ε, κόστος. Εκτός βεβαίως αν το έχει κάνει με, με δόλο. Οπότε εντάξει, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Αλλά το ερώτημα ποια διαδικαστικά σφάλματα είναι αυτά που θα πρέπει να καταγράφονται ίσως ε, ως ε, ε, απλά διαδικαστικά λάθη με μειωμένη επίπτωση στα οικονομικά. Αυτό θα πρέπει να το δούμε ίσως πιο ίσως λεπτομερέστερα. Ευχαριστώ. Κύριε κυρία, Κύριε. έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Εγώ είμαι νέο μέρος στο Κοινοβούλιο από πέρσι ε, στο παρελθόν όμως ήμουν αυτοδιοικητική στο Δήμο της Πράγας. Ε, ε, εργάστηκα επί σειρά ετών στην Τσεχική Δημοκρατία και πρέπει να σας πω και ομολογώ ότι είναι σχετικά νέα όλα αυτά για μένα που συζητούμε εδώ. Αυτή η αρχή του ανεκτού κινδύνου σφάλματος είναι κάτι το οποίο δεν δέχομαι από την αρχή την ίδια. Δηλαδή ούτε επί της αρχής δεν το δέχομαι. Ας πούμε, εγώ ήμουν μέλος ε, στην Επιτροπή Οικονομικών του Δήμου της Πράγας, επαναλαμβάνω, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Καλά, τώρα εδώ δεν είναι τοπική αυτοδιοίκηση, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. <laughs> Ε, αλλά θέλω να σας δώσω αυτή την ε, ε, ιδέα από ένα άλλο πρίσμα. Και ποια είναι τα κριτήρια, πώς ορίζεται δηλαδή αυτός ο ανεκτός κίνδυνος φάρμακος. Αν καταλαβαίνω σωστά τη συζήτηση που γίνεται τώρα εδώ, πρέπει να σας πω ότι έχω κάποιες επιφυλάξεις για τα κριτήρια. Αφενός, δεν έχω κανένα πρόβλημα το ελεκτικό συνέδριο στις εκθέσεις του να χρησιμοποιεί αυτούς τους όρους και τις έννοιες. Αλλά από την άλλη πάλι δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να το έχουμε ως κριτήριο στα προγράμματά μας και να το μετράμε. Γιατί αυτό δίνει ένα θετικό μήνυμα σε εκείνους που δεν είναι πρόθεμοι ε, πάντα να τηρούν τους κανόνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον εισηγητή και για τη συζήτηση που γίνεται, γιατί επαναλαμβάνω για μένα ένα θέμα πρωτόγνωρο και ε, με προβληματίζει και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα από την αρχή της θητείας, αλλά πρέπει να σας πω με εκπλήσει και ιδιαίτερα. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και πάλι για την έκκληση που απευθύνει στα κράτη-μέλη στο κείμενό του. Συμφωνώ. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Κύριε Σάλτεμος. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ελεκτικό Συνέδριο και τον εισηγητή για αυτά που μας είπαν είναι πολύ σημαντική συζήτηση αυτή που διεξάγεται εδώ. Πολύ δύσκολο να γνωρίζουμε ποια είναι η απάντηση. Κάποιοι λέγουν αυτό που κάνουν κάποια κράτη-μέλη δεν αρκεί. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου τα προβλήματα είναι σοβαρότερα από αλλού. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε επί του στόχου μας και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η μείωση των σφαλμάτων, να ελαχιστοποιηθούν τα σφάλματα. Το μηδενικό ποσοστό είναι ανέφικτο βέβαια, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε για να καταλήξουμε στο χαμηλότερο ποσοστό σφαλμάτων που είναι δυνατόν. Γι' αυτό το λόγο είναι δύσκολη η συζήτηση, διότι αν μιλούμε για αποδεκτό επίπεδο ελέγχου, κυρίως στις μικρές χώρες από τις οποίες προέρχομαι και εγώ, από τη Δανία, δημιουργείται η εντύπωση ότι δεχόμαστε αρκετά σφάλματα. Και πιστεύοντας αυτό, προσπαθούν κάποιοι να κρυφτούν και πιστεύουν ότι αυτοί που κρύβονται και που είναι ένοχοι σφαλμάτων μπορούν να κρυφτούν και να μην ανακαλυφθούν. και αυτοί που τα καταφέρουν καλά ανακαλύπτονται. Πρέπει λοιπόν το μήνυμα που θα στείλουμε να είναι σαφές. Θα πρέπει στο βαθμό του δυνατού να ελαχιστοποιήσουμε τα σφάλματα. Δεν πρέπει να συζητούμε όμως μόνο τα σφάλματα, αλλά και τα αποτελέσματα, τα προγράμματα. Ποια είναι τα αποτελεσμάτων των διαφόρων προγραμμάτων. Και αυτό θα πρέπει να μελετηθεί. Έτσι θα πετύχουμε πιο ισορροπημένη λύση. Προς τον εισηγητή θα έλεγα το εξή. Αυτή η ιδέα μιας εναλλακτικής λύσεως είναι έξοχη. Δηλαδή, να πάρουμε τους διάφορους τομείς πολιτικών και να τους εξετάσουμε, αλλά να γνωρίσουμε επίσης να δούμε και ποια είναι η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Διότι αυτό έχει αποφασιστική σημασία. Θέλουμε να βρούμε λύση. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε κάποιον συγκεκριμένα. Θέλουμε να βρούμε μια λύση. Λύση που θα επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων. Λοιπόν, η πρότασή σας ήταν πάρα πολύ καλή, ήταν εξαιρετική. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να Νομίζω ότι πρέπει να ορίσουμε πιο συγκεκριμένα τους όρους που χρησιμοποιούμε. Εδώ στα έγγραφα γίνεται ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ του ανεκτού κινδύνου σφάλματος και του ανεκτού επίπεδου κινδύνου. Τώρα, κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι στην ε, πολιτική συνοχή που την αναφέρουμε συχνά είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε τους δικαιούχους ώστε να εμπλακούν και να ξεκινήσουν ε, καινοτόμες δραστηριότητε. Δραστηριότητε που ίσω ε, να, ε, πρέπει να ξεκινήσουν και μέσω πιλωτικών προγραμμάτων ή κάποιων πειραματισμών. Αν, θέλουν απλώς να κάνουμε, αν θέλουμε να κάνουν απλώ αυτό, τότε το επίπεδο κινδύνου που θα πρέπει να επιτρέψουμε θα πρέπει να είναι πιο ε, υψηλό, εάν θέλουμε η, η πολιτική συνοχή να βασίζεται σε καινοτόμε δραστηριότητε, σε καινοτόμα προγράμματα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το επίπεδο κινδύνου θα πρέπει να είναι πιο υψηλό. Οπότε, σήμερα τι λέμε. ότι αυτή η έννοια του ανεκτού κινδύνου ασφάλματος και του ανεκτού επίπεδου κινδύνου πρέπει να έχει και κάποιο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος που θέλουν να εκπληρώσουν αυτοί οι δύο ορισμοί. Θέλουμε αυτοί οι ορισμοί να χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή προγραμμάτων. Θέλουμε να ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη για τους δύο αυτούς όρους. ώστε να συνεχιστεί η εφαρμογή των προγραμμάτων, είναι απλώς κάτι ενημερωτικό που θα χρησιμοποιηθεί για να αξιολογηθεί εκ των υστέρων η πολιτική μας. Ίσως θα μπορούσαμε να δούμε πού έχει εφαρμοστεί η πολιτική σωστά και πού λανθασμένα, να κάνουμε δηλαδή στον ε, εκ των υστέρων έλεγχο μια αναφορά και να πούμε ότι ίσως το επίπεδο κινδύνου ήταν πιο υψηλό. Και ερωτώ, χρειάζονται αυτές οι κατηγορίες για να, ε, για να ξεκινήσουν να προετοιμάζονται κάποιες κατηγορίες εκ των προτέρων ή χρειαζόμαστε αυτές τις κατηγορίες για να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο εκ των υστέρων. Γιατί στα έγγραφα υπάρχει και μια τρίτη, ε, ένας τρίτος όρος, το κόστος ελέγχου που σημαίνει ότι αν θέλουμε να ελέγξουμε περισσότερο για να έχουμε λιγότερα λάθη, αυτό σημαίνει ότι το κόστος ελέγχου θα είναι υψηλότερο. Οπότε, τελικά ο ρόλος ο δικός μας ποιος είναι. Πού είναι η ισορροπία, ποιο είναι το σημείο ισορροπίας μεταξύ των δύο. Θέλουμε να αυξήσουμε το κόστος ελέγχου στο άπειρο για να, βρούμε, να έχουμε τελικά καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να βρούμε αυτό το μαγικό σημείο ισορροπίας το οποίο θα μπορούσε να είναι αποδεκτό από όλους εάν θέλουμε να έχουμε καινοτόμε και θαραλές δραστηριότητες. Αν ναι, τότε πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι θα υπάρχει πάντα ένα περιθώριο λάθος. Γι' αυτό πρέπει σαφώς να ορίσουμε τι είναι ο ανεκτός ε, κίνδυνος σφάλματος Χρειαζόμαστε αυτό τον ε, όρο για να ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη για το τι επίπεδο κινδύνου θα δεχτούμε. Ίσως να δεν έχουν απάντηση όλες αυτές οι ερωτήσεις, γιατί εκ των προτέρων δεν μπορούμε να πούμε ποιο θα είναι το, επίπεδο ανεκτού, το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Θέλουμε να ενισχύσουμε, να αυξήσουμε το, το, το κόστος ελέγχου ε, όσο πάει, απλώς για το είναι σκόπιμο πολιτικά αυτό. Ο κύριος Σοντή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως και άλλους συναδέλφους, με ενοχλεί και εμένα λίγο η σημερινή συζήτηση. Δηλαδή αισθάνομαι άβολα να βγω να πω ε, στους ε, πολίτες για το, ότι συζητάμε για το αν θεχόμαστε ή όχι σφάλματα. Ε, έχουμε συλλογική ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ε, και το ελεκτικό συνέδριο ε, με το συμπάθειο. Πρώτον υπάρχει ο εξής κίνδυνος που ελοχεύει. Να συγχέουμε το κατόφλι σημασίας με τον κίνδυνο του ανεκτού σφάλματος. το κατόφλι σημασίας αξιολογείται στον οικονομικό έλεγχο. Ε, μας δίνει το ελεκτικό συνέδριο μια έκθεση. Εμείς κάνουμε ε, ό,τι θεωρούμε σκόπιμο. Δίνουμε απαλλαγή ή όχι. Και εδώ είναι ένας πρώτος κίνδυνος. Γιατί καμιά φορά διαβάζοντας τα έγγραφα και με τη ερμηνεία θα πρέπει να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στον κίνδυνο και στο κατόφλι της σημασίας ή της ασημαντότητας ε, της στατιστικής. Ε, μετά γίνεται λόγος για το κόστος των ελέγχων, ότι είναι ακριβή η έλεγχη και χρειάζεται προσοχή. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να θέσω επιτάπητος κάτι άλλο. Ε, να κάνω μια πρόταση, Πρόεδρε, στην Επιτροπή μας να μπει και μια άλλη παράμετρος που είναι το κόστος της δικής μας οργάνωσης. Γιατί ε, μπορεί να είναι αυξημένο το κόστος των ελέγχων, αλλά για ποιο λόγο είναι αυτό αυξημένο. Διότι είναι περίπλοκη η οργάνωσή μας. Γιατί κάθε φορά λέγουμε ότι γίνονται σφάλματα διότι είναι περίπλοκη νομοθεσία. Μα δεν είναι μόνο η νομοθεσία περίπλοκη και ο τρόπος που οργανωνόμαστε οι ίδιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Εγώ με. πώς κάνεις εσωτερικό οικονομικό έλεγχο σε εξωτερικές δομές. Τα κράτη-μέλη είναι κυρίαρχα. Πώς κάνεις εσωτερικό έλεγχο σε κυρίαρχα κράτη. Και ποιος μπορεί να με διαβεβαιώσει ότι οι αρχές ελεγκτικές των κρατών είναι ανεξάρτητες. Το είπε και ο Επίτροπος αυτό. Εγώ πήγα ε, να δω τις ελεγκτικές αρχές στους Γάλλους ορκωτούς ε, λογιστές και τους ρώτησα ποιος ορίζει ε, την αμοιβή σα, Ποιό σα διορίζει, ο υπουργό. Ε, είναι αυτή η ανεξάρτητη τότε. Δηλαδή η οργάνωση ε, του συνόλου και συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατών Μελών ε, αξίζει τον κόπο να μετρηθεί. Πόσο κοστίζει η οργάνωση αυτή για τη συνυπευθυνότητα κυρίως γιατί είναι τα προβλήματα για τη διαχείριση των κονδυλίων και γιατί έχουμε προβλήματα με τα κάποια κράτη-μέλη. Βεβαίως λόγω του περιπλόκου αλλά και λόγω ε, της διοικητικής μηχανής που ασχολείται. Στο παρελθόν είχα ε, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκεφτεί να δημιουργήσει τη δική τη οικονομική διαχείριση. Ένα σώμα. Ε, δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα, δεν έχει έρθει. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να πούμε πόσο θα κόστιζε μια οικονομική διακυβέρνηση, διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο σήμερα κοστίζει αυτή. Βεβαίω είναι περίπλοκη η διαχείριση αλλά και η οργάνωση μας επαναλαμβάνω. Τα κράτη-μέλη λένε θέλω τα λεφτά μου πίσω. Ε, εντάξει, γιατί ε, αυτοί διαχειρίζονται. Δεν θα μπορούσαμε εμείς όμως να εξευρωπαίσουμε τρόπο τεινά τα, τη διαχείριση και να τα διαχειριζόμαστε εμείς. για να γίνονται έλεγχοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιο φθηνοί, θέλετε. Διότι ο Κεντρικό έλεγχο, φαίνεται, φαίνεται λέω, χρειάζεται μελέτη. Πιο φθηνό και με λιγότερους κινδύνου και με λιγότερα σφάλματα. Λοιπόν, ε, να πούμε ότι είναι περίπλοκα ναι, ε, τα νομοθετικά, αλλά είναι περίπλοκα και τα οργανωτικά στο σύνολό του. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Χατζημαρκάκη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την ε, διευκρίνηση για το ότι τα κράτη-μέλη είναι χειρότερα από την Κομισιόν. Ε, εντάξει, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, τόσο απλά. Σα παραπέμπω στην εξέταση που έκανε το Ελεκτικό Συνέδριο σε ό,τι αφορά τον τομέα τη παιδεία. Εκεί το Ελεκτικό Συνέδριο για 42% των περιπτώσεων διεπίστωσε ε, ένα, ένα ποσοστό λάθους. Και αυτό έχει να κάνει με τι ε, πληρωμέ τη Κομισιόν προς τους δικαιούχους. 42% ε, είναι αρκετά υψηλό, αν δείτε δηλαδή ε, ακριβώς τι έγινε. Εντάξει, ήταν ε, ε, για τα σημασίας λάθη στις, σε 50% των περιπτώσεων δεν θα ήταν και επιλέξιμο το πρόγραμμα για χρηματοδότηση. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο τα κρατημένα είναι χειρότερα από την Κομισιόν. Και κύριε Επίτροπε, ε, θα διαφωνήσω μαζί σας, γιατί εκεί που λέτε ότι ε, είναι δύσκολο το θέμα σε ό,τι αφορά την κατανομή των ε, προμηθών αρμοδιοτήτων για την συνοχή. Αλλά και για την γεωργία είναι ξεχωριστές οι αρμοδιότητες και εκεί τα πράγματα πάνε καλά. Γιατί η Κομισιόν εδώ και πολλά χρόνια κάνει σωστά τη δουλειά της και έχει σαφή συστήματα, δαπανηρά αλλά σαφή συστήματα ελέγχου. Κοστίζουν βεβαίω, είναι δαπανηρά, αλλά έχουν αποτελέσματα. Και μάλιστα είναι πολύ ενθουσιασμένοι όσοι χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα συστήματα ελέγχου, τουλάχιστον στην, στον τομέα τη ε, γεωργία. Επίση, να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και να τον συγχαρώ για την, ε, δραστηριότητα, για την έκθεση των ε, πεπραγμένων, των δραστηριοτήτων. Όντω, οι γενικοί διευθυντέ γνωρίζουν, αναγνωρίζουν ότι γίνονται λάθη και κατονομάζονται τα κράτη-μέλη που υπάρχουν προβλήματα. Οπότε το σέβομαι και, το... και σας ευχαριστώ. Γιατί αυτό δείχνει ότι αναπτύσσονται τα συστήματα και βελτιώνονται από χρόνο σε χρόνο. Και χαίρομαι, αναφέρατε και τα αριθμητικά στοιχεία, που μιλήσατε για το ε, σύστημα της ε, αναστολής ή της παύσης και το χρησιμοποιείτε. Μιλήσατε για 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία ε, ανεστάλησαν. Και για το 2.000 ε, ευρώ μιλήσατε για 15 αποφάσει για τέτοιε αναστολέ. Για το 2010 περίπου διπλάσιο ο αριθμό, όπω είπατε. Αυτά είναι καλά αριθμητικά στοιχεία. Είναι εξαιρετική λοιπόν η δουλειά και χαίρομαι που λειτουργεί το σύστημα. Και στον ιστορικό έλεγχο βεβαίω, ε, εκπαίδευση, έρευνα και εκεί θα πρέπει να γίνει κάποια βελτίωση. Τώρα, είπατε, κύριε Επίτροπε, και το αναφέρατε και με νούμερα, ότι το σύστημα αυτό είναι πολύ δαπανηρό. Το είπε και ο κύριο Σοντή ε, για τον ε, τομέα με ενέργεια και μεταφορές και έρευνα. Αναφέρατε κάποια αριθμητικά στοιχεία για ένα επιπλέον ελεγκτικό σύστημα που μιλήσατε για επιπλέον 90 ε, έως 150 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μείνουμε κάτω από το 2% περιθώριο λάθους. Έτσι το κατάλαβα εγώ, αυτό που είπατε. Το σημειώνω, αλλά πρέπει να σας πω ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, βρήκε στο κεφαλαίο 1.44 ότι μέχρι τώρα τα, τα, τα επιστραφέντα ε, κονδύλια για την, ε, για την συνοχή, για τις διορθώσεις, μιλούμε για 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Αν τα συνυπολογίσουμε όλα, είναι προφανώς περισσότερα, και μιλούμε για 476 ε, εκατομμύρια που, επανα, που ε, επανήλθαν, δηλαδή 20%. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να επενδύσουμε περισσότερο σε καλύτερα ε, συστήματα ελέγχου, ώστε να λαμβάνουμε κάθε φορά τέτοια μεγάλα ποσά ε, ως επιστροφή. Και ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε έτσι μια εικόνα και για το σύνολο του ελεγκτικού συστήματος. Γιατί είπατε για 90 150 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Αλλά μιλούμε μόνο για την έρευνα, τι μεταφορές και την ενέργεια. Αν έχουμε ένα εξίσου υψηλής ποιότητας ελεγκτικό σύστημα για τη γεωργία, όπως έχουμε για τη γεωργία, σε όλου του τομεί πόσο θα, πόσο θα κόστιζε. Θα πρέπει να το δούμε ίσω. Αξίζει τον κόπο. Αν δούμε δηλαδή και πόσα χρήματα έχετε δαπανίσει και που δεν έχετε ζητήσει ε, όσα χρεώσετε ως καταφληθέντα. Για την κυρία Γιάλα Σέντερ δεν θέλω, να, δεν θέλω να την ξαναπροσβάλλω, οπότε δεν θα πω τίποτα. Ε, αλλά μιλήσαμε για τα σταλίες και έτσι και στο μυαλό μου μπορώ εύκολα να υπολογίσω πόσα είναι τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά αν είναι τα νούμερα τόσο υψηλά, νομίζω ότι πρέπει να το λέμε. Εγώ δεν προσπαθώ να προσβάλλω κανέναν εδώ. Ούτε θέλω να καταδείξω ποιο είναι ο καλό και ποιο είναι ο κακό. Αλλά ε, το κάνω για να γίνουμε εμεί οι ίδιοι καλύτεροι. Βεβαίω η χειρότερη κατάσταση ε, κατά κεφαλή είναι, στην, είναι η Ελλάδα, έτσι. Αλλά η Ελλάδα επιστρέφει και περισσότερα όταν διαπιστώνονται λάθη. Με απόσταση, δηλαδή η παρασάγκα απέχει από όλου του υπόλοιπου η Ελλάδα. Χάρηκα κύριε Ολμπριχτ που μιλήσατε για καινοτόμα προγράμματα. Τα καινοτόμα προγράμματα όντω ζητούνται περισσότερο από ποτέ. Και βεβαίω πρέπει και πάλι να ε, επενέσω την ε, Κομισιόν, γιατί κύριε Σεμέτα με τους, ε, με τους συναδέλφους σας ε, συζητήσατε για το πώς μπορούμε στο μέλλον να λειτουργήσει καλύτερα ο τομέας της συνοχής και το παρουσιάσατε. Και εσείς μιλήσατε για ένα καινοτόμο εργαλείο, για τα μπόνους. Δηλαδή δεν, δεν προωθούμε, δεν, δεν χρηματοδοτούμε από την αρχή, αλλά όταν βλέπουμε μία βελτίωση στην, στην πολιτική ας πούμε απασχόλησης, τώρα, τότε παίρνει μπόνους. Αυτό νομίζω ότι είναι εξαιρετική πρόταση για τον τομέα της πολιτικής έρευνας αυτή την, αυτή την, ε, αυτό, αυτό το, αυτή την προσέγγιση θα την, ε, θα τη χρησιμοποιήσουμε. Γιατί από την αρχή δεν μπορεί κανείς να χρηματοδοτήσει την έρευνα. Για την έρευνα λοιπόν και την καινοτομία, αυτό που όντως είναι καινοτόμο και που δίνει καινούργιε ιδέες στην αγορά, μπορούμε να το, το επιβραβεύσουμε με ένα μπόνους. Και εκεί είναι και η κατάχρηση μικρότερη και τα λάθη θα είναι επίση, τα σφάλματα θα είναι επίση λιγότερα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα είναι μια αλλαγή του συστήματο για την οποία θα πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω, Επίτροπε Σεμέτα. Και κλείνοντα. να κάνω μια παρατήρηση σε σχέση με αυτό που είπε η συνάδελφο ε, Σάλντε Μοζή. Ε, αυτή η προσέγγιση που προτείνετε εσεί, ε, δηλαδή το ανεκτό επίπεδο κινδύνου, δεν θα πρέπει να το δούμε σαν ένα πέπλο το οποίο χρησιμοποιούμε εμείς για να, πούμε, να χρυσώσουμε το χάπι στους πολίτες. Σε όλες τις πολιτικές ομάδες βλέπετε ότι υπάρχουν έτσι, ε, ε, υπάρχει ε, δισταγμός και ακόμη και το ελεγκτικό συνέδριο είναι, το ελεγκτικό συνέδριο είναι αυτό που εισήγαγε αυτό τον όρο το, το 2004 και πάλι υπήρχε πρόβλημα στον οριστή σαφώ αυτό ο όρο. Οπότε α είμαστε έτσι λίγο συγκρατημένοι με την εφορία που δημιουργείται. Ε, στην, στο κοινοβούλιο δεν είναι τόσο ευτυχή τα πράγματα, θα το παρατηρήσετε και από τη συζήτηση. Και δεν έχουμε και δεν είμαστε και πεπισμένοι κι εμείς από, από, την, από τον όρο αυτό. Οπότε πρέπει να, να δούμε και τι ακριβώς λέμε τελικά στους φορολογούμενους. Λέμε, τι λέμε προς τα έξω. Νομίζω ότι θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να γίνουμε καλύτεροι, να εργαστούμε πιο, πιο αυστηρά, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, να έχουμε καλύτερους, ε, καλύτερα συστήματα ελεγκτικά, παρά να, να ανακυκλώνουμε συνέχεια κάποιες φιλοσοφικές ιδέες που ουσιαστικά στο τέλος είναι αυτό που κάνουμε, αυτό που κάνουμε μετατρέπεται σε, ένα, σε μια, ένα και καλυμμένη, μια και καλυμμένη πολιτική. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει από την κυρία Γκαλουλάιτε, την εκπρόσωπο του Ελεκτικού Συνεδρίου, κάποιο σχόλιο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση. Πρώτα απ' όλα να αναφέρω την απλούστευση Ακούσαμε ότι η απλούστευση θα μπορούσε να οδηγήσει και σε ένα εργαλείο που βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και σε συστήματα που ανέχονται περισσότερο τον κίνδυνο. Είμαστε σίγουροι, η απλούστευση αφορά την περικοπή τη μη απαραίτητη ή άσχετη γραφειοκρατία για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων. Θα είναι πιο κομψό το σύστημα, όπου θα γίνονται λιγότερα σφάλματα, διότι υπάρχουν λιγότεροι κανόνε, επίσημοι και τυπικοί κανόνε. Αυτό αφορά την απλούστευση. Ο κ. Σοντή σωστά είπε ότι τα προγράμματα μπορούν να ανασχεδιαστούν αν έχουμε από απλούστευση και περικοπή γραφειοκρατία και βλέπουμε ότι η διαχείριση παραμένει περίπλοκη, ίσως θα πρέπει να ξανασχεδιάσουμε την προσέγγιση ριζοσπαστικά. Τρίτη επιλογή, θα υπάρχει κάποτε, να σταματάει μια δραστηριότητα αν τίποτα δεν οδηγεί σε λύση. Και μόνο εάν έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν διερευνηθεί τα πάντα για την επίτευξη του στόχου και ο κίνδυνος εξακολουθεί να είναι υψηλό, τότε θα έπρεπε να συζητούμε το ανεκτό επίπεδο σφάλματος. Και όταν συζητούμε το ανεκτό επίπεδο σφάλματος, πέραν από τον επαναλαμβανόμενο κίνδυνο, υπάρχει και ο κίνδυνος της διαχείρισης. Ποιος είναι αυτός? Αν πάρει ξεχωριστό δείγμα για τη συνοχή. Δεν δημιουργούν όλοι τα σφάλματα. Το 1 τρίτο από τους ελεγχομένους μόνο δημιουργεί τα περισσότερα σφάλματα. Άρα, αν ανακοινωθεί στόχος υψηλότερος από το στόχο του ελεκτικού συνεδρίου εκείνοι που δεν έκαναν σφάλματα ίσως να τίνουν να μειώσουν το επίπεδο ελέγχων και το κόστος των ελέγχων και εκείνοι που κάνουν περισσότερα σφάλματα ίσως να μην πετύχουν τους στόχους. Άρα τελικά το πρόβλημα διαχείρισης ίσως να καταλήξει να είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο Επίτροπος, ο κ. Σαμέτα, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Συμφωνώ απολύτως με τον εισηγητή. Ε, ως προς το γεγονός ότι η ίδια η έννοια του ανεκτού κινδύνου σφάλματος δεν είναι εύκολη και ε, σαφής υπόθεση. Οι υπηρεσίες μου είναι στη διάθεσή σας για να σας εξηγήσουν τον ορισμό και την έννοια που κρύβεται πίσω από τις προτάσεις μας. Θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα είπε ο κύριος Οντί. Και πολύ σωστά ε, τόνισε το ζητήμα. Αυτό είναι ε, μια, είναι ένας ορισμός που χρησιμοποιείται στη διαχείριση, στο management. Ε, κάπου πρέπει να βάλει ορόσημα όταν διοικείς, διαχειρίζεις ένα σύστημα για να προσανατολίζεις τη δράση σου για να φτάσεις σε αυτούς τους στόχους. Αυτό κάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό προτείνει. Δεν αναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αποφασίσει αυτό, αλλά σε εκείνους που αποφασίζουν και παίρνουν τις οικονομικές αποφάσεις για να πούνε ποιο είναι το επίπεδο κινδύνου και ποιο είναι το ανεκτό και το ανεκτό κίνδυνο ή το, ποιο είναι το ανεκτό επίπεδο σφάλματος που είναι ελαφρώς διαφορετικές έννοιες και εντός της έννοιας του ε, ανεκτού κινδύνου σφάλματος όταν διαπιστώνεται οποιοδήποτε σφάλμα θα πρέπει αυτό να διορθώνεται και να ανακτώνται τα κονδύλια. Uh, είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να κατανοούμε πώς λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Εγώ είμαι πολύ μεγάλος οπαδός και υποστηρικτής της απλούστευσης, αλλά πάντα θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι για να γίνουν οι απλοποίησεις χρειάζεται χρόνος. Εγώ είμαι προσιλωμένος σε αυτή την υπόθεση και οι συνάδελφοι ε, επίτροποι για την επόμενη γενιά προγραμμάτων να προτείνουμε όποιες απλουστεύσεις χωράνε. Αλλά αυτό σημαίνει θα ξεκινήσουμε από το 2014 και μετά. Και η απαλλαγή θα έρθει το 2016, ίσως και αργότερα για τα έτη αυτά. Οπότε θα πρέπει να ασχοληθούμε και με την παρούσα κατάσταση, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τώρα το, πρόγραμμα, το πρόβλημα. Και η έννοια αυτή ε, είναι μία από τις απαντήσεις και δίνει και αντικειμενικά κριτήρια στην αρχή που χορηγεί την απαλλαγή για τον τρόπο με τον οποίο ε, εργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς είναι οι ελεγκτικοί της μηχανισμοί και πώς μπορούν να αξιολογούνται. Ο κύριος Γκάιερ είπε ότι είναι σημαντικό να συμμετέχει και το Συμβούλιο στη συζήτηση αυτή. Και ειλικρινά και η δική μου προσέγγιση αυτή είναι και η δική μας πρόθεση. Να συζητήσουμε αυτό το θέμα και με το Συμβούλιο. Γιατί όχι και στον τριμερή διάλογο γιατί είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο το Κοινοβούλιο, ε, αλλά και το Συμβούλιο που έχει λόγο για αυτά τα θέματα. Και έρχομαι στις ε, εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας οικονομικής διαχείρισης και ε, προωθεί την έννοια αυτή πάρα πολύ σοβαρά ο εισηγητής. Εδώ έχω να σας πω τα εξής δύο. Έχω δύο παραδείγματα. Ε, μία μόνο δήλωση έχει υπογραφεί ε, από τον Υπουργό και έχει υποστεί έλεγχο από τον, τον συνέδριο της χώρας. Και το θέμα είναι ότι ε, ε, το επίπεδο σφάλματος ε, και σε αυτές τις χώρες είναι υψηλότερο από εκείνο που αξιολογεί το ελεκτικό συνέδριο. Ενώ ότι ακόμα και αν έχουμε υπογραμμένες τις δηλώσεις αξιοπιστές των κρατών μελών, αυτό δεν λύνει όλα μας τα προβλήματα. Και, όπως είπε η κυρία Γιάλα, έχουμε και ομοσπονδιακά κράτη. το ξέρω πολύ καλά και ο εισηγητής αυτό που προέρχεται από μια ομοσπονδιακή χώρα. Και είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι ένας ομοσπονδιακός υπουργός θα βάλει την υπογραφή του για δήλωση διαχείρισης και αξιοπιστίας ε, που θα έχουν υποβάλει κάποιοι υφιστάμενοι υπουργοί του ε, οικονομικών ε, των κρατηδίων. Δεν ξέρω τις νομικές λεπτομέρειες βέβαια στη Γερμανία, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να θεωρείται αυτό μέχρι και αντισαγματικό. Υποθέτω, λέω, δεν, δεν το λέω με βεβαιότητα αυτό. Εσείς τι προτείνετε τώρα να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να μας φέρνουν δηλώσεις αξιοπιστίας από το σωστό επίπεδο. Δηλαδή ο, ο ύπατος διαχειριστής που πραγματικά διαχειρίζεται τα κονδύλια αυτά να δίνει την υπογραφή του και τη βεβαίωσή του ότι είναι όλα εντάξει. Βάσει ε, των αρχών της χρηστής διαχείρισης. Αυτό το σύστημα το εφαρμόζουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από ό,τι φαίνεται λειτουργεί. Σωστά. Και εσείς ο ίδιος χειροκροτήσατε, καλωσορίσατε την ετήσια έκθεση πεπραγμένων ή δραστηριοτήτων ε, που ακολουθεί αυτό το σύστημα και προτείνουμε να το επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς δαπανών και κατά τα άλλα και ειρήστον στη Γεωργία αυτό ήδη ισχύει. Και θα θέλαμε να μεταφέρουμε την εμπειρία αυτή και αλλού και σε άλλους τομείς ε, πολιτικής και πιστεύουμε ότι θα φέρει καλά αποτελέσματα. να μπω λίγο σε κάποιες λεπτομέρειες. Αναφερθήκατε στα δικά μου στοιχεία, στα νούμερα, για το επιπλέον κόστος ελέγχου που ανέφερα και εγώ στην παρουσίασή μου. Και οι υπολογισμοί δικοί μας αποδεικνύουν ότι αν θέλουμε να φύγουμε από το 3% και να πάμε στο 2% επίπεδο σφάλματος στην έρευνα, αυτό θα σήμαινε κόστος από 90 εκατομμύρια ευρώ 150 πλέον. Γιατί, ενώ ε, η ανάκτηση από αυτό το 1% θα ήταν μόλις 72 εκατομμύρια. Δηλαδή θα κόστησε περισσότερο ο έλεγχος παρά η ίσπραξη και ε, περισσότερος έλεγχος σημαίνει περισσότερο φόρτο ε, στους ώμους των δικαιούχων. Βεβαίως υπάρχουν και ε, ε τεχνικές, το είπε και ο κύριος Σοντή αυτό, για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Ε, το βασικό μέτρο είναι να αυξηθούν οι έλεγχοι σε επίπεδο δικαιούχων και το είπε αυτό και το ελεκτικό συνέδριο. Uh, και ε, στην έκθεσή του. Και αυτό σημαίνει επιπλέον ε, βάρος προφανώς και επιβράδυνση της εφαρμογής των προγραμμάτων και άλλες ανητικές συνέπειες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να βρούμε ε, μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα ελέγχων και την αποτελεσματικότητά τους πάντα, τι δηλαδή, επιδιώκουμε και να πιάνουν τόπο και τα κονδύλια. κάτι άλλο που είναι επίσης σημαντικό υπόθηκε ότι φέρουν τα κράτη-μέλη στην εφαρμογή. Αν συμφωνήσουμε για το ανοιχτό κίνδυνο σφάλματος ως προς την έννοια έτσι και το επίπεδο του, αυτό θα έβρισκε εφαρμογή όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και στα κράτη-μέλη που διαχειρίζονται έτσι, στη συνυπευθυνότητα κονδύλια μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουν και με πολλά λάθη και σε ψηλό επίπεδο πούμε, σε ποσοστό θα πρέπει να μειωθεί αυτό έτσι ώστε να ε, φτάσουν στο επιθυμητό ορόσημο, το benchmark. Και αν θέλετε μπορούμε να κατονομάζουμε και να διαπομπεύουμε και κράτη-μέλη που δεν ε, φτάνουν σε αυτό το στόχο γιατί έχουμε πλέον εισαγάγει ένα αντικειμενικό κριτήριο και εκεί μπορούν να κρίνονται τα κράτη-μέλη εκ του αποτελέσματο. ότι ο ένα θα πάει καλύτερα, ο θα πάει χειρότερα. Uh, uh, Αυτά. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα σημεία που σας απασχολούν και ε, αναφέρατε κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Συμφωνώ με τον κύριο Γκάιερ που είπε ότι θα μπορούσαμε να δούμε πώς θα διευρύνουμε αυτή την έννοια ενδεχομένω. Βεβαίως, ο είναι τέλειος και πάντα χωρούν βελτιώσεις. Μπορούμε πάντα να το κάνουμε αυτό και να συζητούμε και με το Συμβούλιο. Λοιπόν, Προσβλέπω στη συνέχιση της συζήτησης αυτής και στη συνεργασία μας θα ενημερώσουμε και το Συμβούλιο και άλλους ενδιαφερομένους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα ζήτησε να μιλήσει. Ναι, Πρόεδρε. Ζήτησα το λόγο για να ζητήσω κάτι από εσά. Θα σας παρακαλούσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας στείλει όλη την πληροφόρηση που έχει για αυτή την περίπτωση ε, της ε, υπογεγραμμένης δήλωσης αξιοπιστία. Χρόνια ολόκληρα το κυνηγάμε αυτό το θέμα, σαν να ήταν το Άγιο Δισκοπότηρο. Ο Τέρι Γουίν, παλιός μας συνάδελφος, το είχε ξεκινήσει και βλέπουμε ότι μια χώρα που το εφαρμόζει μετά τρέχει και δεν φτάνει. Αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, δυσεπίλητα και άλλη τα τελικά. Ε, να μην συνεχίζουμε τώρα να ε, τροφοδοτούμε διάφορους μύθους εδώ πέρα και άπιαστα όνειρα που μας δυσκολεύουν την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ε, συμφωνώ με την πρόταση της κυρίας Αγιάλα. Θα ήθελα και εγώ βάσει τον όσον είπε ο εισηγητής και αυτά που είπε η κυρία Αγιάλα και ο συνάδελφος Οντί. Έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα πρέπει να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε πού υπάρχουν οι συγκρούσεις συμφερόντων. Και εκείνοι που θα πρέπει να ελέγξουν πολύ συχνά συνδέονται ε, με εκείνους που κάνουν χρηματοδότηση ή τους δικαιούχους. Αυτή είναι αφηρημένη έννοια, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις το είδαμε και μπροστά μας. Όπως στη χώρα μου, στην Ιταλία, που καμιά φορά η κατάσταση δεν είναι καθόλου θετική. Και άλλη μια πτυχή, κάτι που συμβαίνει συχνά. Εκείνος που θέλει να πάρει τους πόρους, να πόρους με αθέμητο τρόπο ή θέλει να εξαπατήσει, ξέρει να κινηθεί με τέτοιο τρόπο που τυπικά τα πάντα είναι μια χαρά. Όσον αφορά τους τύπους, τις νομικές διαδικασίες, τα πάντα είναι στη θέση τους. Αυτό σημαίνει ότι η έλεγχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικη όσον αφορά την ουσία. Μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά παραδείγματα. Κάποια φορά, θυμάμαι, υπήρχε μια εταιρεία που είχε πάρει 4 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματοδοτήσει ευρωπαϊκέ στην Ιταλία για να κάνει DVD και CD. Επίσημα, τυπικά όλα ήταν καλά. Εκείνη η επιχείρηση τα έκανε τα πάντα εκτός από τα DVD και τα CD. Η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ξέρουμε ότι είναι σημαντική έλεγχη και δαπανηρή και θέλουμε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με το κύριο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ε, διάλων άλλων φορέων όπως είναι το Ελεγχτικό συνέδριο και τα εθνικά Ελεγχτικά συνέδρια να δούμε πώς μπορεί να συνεργαστούν όλοι με τους διάφορους φορείς σε εθνικό επίπεδο που ασχολούνται με τους ελέγχους της νομιμότητας και από αυτή τη σκοπιά και στο μέλλον ίσως η Όλαφ μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτά που έκανε κατά το παρελθόν. Θέλω να σε ευχαριστήσω όλους, ιδιαίτερα τον εισηγητή, διότι ήταν πάρα πολύ καρποφόρα αυτή η προσπάθεια και δουλειά. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, μπορούμε να πάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης, που αφορά μια μελέτη με θέμα τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΜΚΟ, και χρηματοδότηση αυτών μέσω από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ο κ. Χέλνερ δεν είναι εδώ, ο εισηγητής που αντικαθίσταται άριστα από τον συνάδελφο Ήταλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφός μας, ο κ. Χέλνερ, είναι αλλού γιατί έχει επαγγελματικέ επαγγελματικές υποχρεώσεις. Προσπαθήσω να το αντικαταστήσω. έκανε έξαχη δουλειά, παρουσίασε μια ολόκληρη σειρά συμπερασμάτων που θα ήθελα να παρουσιάσω. Το θέμα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Είναι καλό να διεξαχθεί μια συζήτηση όσον αφορά τα διάφορα σημεία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν περίπου 3.000 μη κυβερνητικέ οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1,4 εκατομμύρια ευρώ το 2010. Πολλά χρήματα ε, και πολλές με κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ωφεληθεί από αυτή την ε, χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να επικαιροποιήσει τη στρατηγική της και τους ορισμούς της. Ξέρετε ότι κάθε γενική διεύθυνση μπορεί να καθορίσει ως φρονή καλύτερο τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση και τι δεν είναι. Δεν υπάρχει ορισμός, ένας ενίος και αποκλειστικός ε, ορισμός του τι αποτελεί μια μη κυβερνητική οργάνωση. Άρα ίσως θα πρέπει να το αποφασίσουμε αυτό, να έχουμε έναν ορισμό. Κάθε φορά κινδυνεύουμε να καταλήξουμε σε κάποιους ορισμούς που είναι πάρα πολύ περιοριστικοί. Χωρίς να λησμονούμε ότι θα πρέπει να υπερασπιστούμε και την ανεξαρτησία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αν ο ορισμός είναι πάρα πολύ περιοριστικός, κινδυνεύουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, να μην είναι πλέον πολύ ανεξάρτητε. Δεν θέλουν να στραφούν προ άλλη χρηματοδότηση, διότι θεωρούν ότι θα μπορεί να επηρεάζεται πολύ από την πολιτική βούληση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε την κατάσταση αυτή, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτεί κάποιε μη κυβερνητικέ οργανώσει, περιμένοντα κάτι σαν ε, αποτέλεσμα, σαν κέρδο. Αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί. Τώρα όσον αφορά τη χρηματοδότηση πάντα. Ίσως θα ήταν καλύτερο να έχουμε μακροχρόνια χρηματοδότηση παρά βραχυπρόθεσμη. Πιο μακροπρόθεσμη. Διότι αν έχουμε βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις, αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την περίπτωση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ε, έχουν υπό τον έλεγχό τους διάφορες άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Θα πρέπει να κάνει συστηματικές αξιολογίες Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των διαφόρων συστημάτων της για τη χρηματοδότηση. Νομίζω ότι έχουμε συλλέξει πληροφορίες από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και σύμφωνα πληροφορίες γνωρίζουμε ότι το σύστημα είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό και χρειάζεται πολλή δρόμος για να πάρουν τη χρηματοδότηση αυτές οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Μάχη ολόκληρη. Να μην λησμονούμε και την διαφάνεια. Πρέπει να δημοσιεύεται ο κατάλογος των ε, δικαιούχων. Σε ιστοσελίδες, στο διαδίκτυο, να μπορούν να παρουσιάζονται οι δικαιούχοι των διαφόρων ε, χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ, παραδείγματο χάρη, να μπορώ να ελέγξω ποιε είναι οι φιλανδικέ μη κυβερνητικέ οργανώσει που έχουν λάβει αυτή τη χρηματοδότηση. Για την ώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αν θέλουμε να εγγυηθούμε την διαφάνεια του συστήματο, θα πρέπει να έχουμε ένα ανεπτυγμένο σύστημα δημοσιεύσεως των δικαιούχων έναν κατάλογο αρκετά λεπτομερή των δικαιούχων των χρηματοδοτήσεων. Ευχαριστώ, λέει ο Προέδρο, τον συνάδελφο τον κύριο Ήταλα. Έχετε το λόγο. Θα αναφερθείτε περισσότερο εργασίε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ήτελε, για τα πρώτα εισαγωγικά σας λόγια για τη μελέτη αυτή. Θα ήθελα σύντομα να σας την παρουσιάσω με τον συνάδελφο Μάικλ Χάμερ από το One World Trust. Από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010 κάναμε τη μελέτη αυτή και μελετήσαμε κυρίως δύο πράγματα. Πριν σας πω για το περιεχόμενο της παρουσίασης, σας μιλήσω για τη μεθοδολογία και τους στόχους για να φτάσουμε σε αυτή. Και μετά ε, ε, θα σας αναφέρω τα βασικά μας ευρήματα και τέλος ε, τις συστάσεις και τα συμπεράσματά μας. Λοιπόν, τι προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Να κοιτάξουμε τα εξής δύο βασικά θέματα. Το πρώτο είναι οι επιδόσεις της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΜΚΟ πόσο καλή είναι η συνεργασία αυτή, πόσο αποδίδει, αν ε, έχει καλά αποτελέσματα και αν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες ε, των διαφερομένων για τη συνεργασία με τις ΜΚΟ και, και επίσης κάτι άλλο που μας απασχόλησε ήταν η διαφάνεια. για τη χρηματοδότηση. και είναι προσβάσιμες αυτές οι πληροφορίες. Έχει ο κόσμος ενημέρωση και χρησιμοποιούν το Μητρό ε, Εκπροσώπων Συμφερόντων οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. we Συνεργαστήκαμε με πολλούς, ε, συναντήσαμε πολλούς γενικούς διευθυντές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γενικό Γραμματέα και τον κύριο Σεύκοβιτς ε, και τις υπηρεσίες του μάλλον τον κύριο Σεύκοβιτς ε, και στα κράτη-μέλη κάναμε επαφέ και είχαμε συνεντεύξει κυρίω στην Ισπανία και τις κάτω και με πολλές μήκυο κάναμε και μια μελέτη, μια έρευνα καλύτερα όπου κοιτάξαμε ποιες είναι οι μη κυβερνητικές ε, οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, ε, την ανθρωπιστική και την παιδεία και την εκπαίδευση. 258 ε, ήταν, 120 από 21 κράτη-μέλη και τέλος κάναμε και κάποιες πιο εμπεριστατωμένες έρευνες και μελέτες για να δούμε πώς Γίνεται η συνεργασία αυτή σε διάφορες γενικές διευθύνσεις πολύ συγκεκριμένες. Μελετήσαμε τη συνεργασία ε, της Ισπανικής Οργάνωσης ε, Υπηρεσίας μάλλον για τη Διεθνή Συνεργασία και ε, το Ολλανδικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πώς συνεργάζονται λοιπόν με ΜΚΟ, ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικές, τι μπορεί να εμπνεύσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ε, συνεργάζεται. Να σας δώσω γενικότερα κάποια στοιχεία, το είπε ο κύριο Σίτελε προηγουμένω, αλλά και προηγουμένω είχαμε καθίσει μαζί στο γραφείο του να κοιτάξουμε τη διαφάνεια για στην οικονομική διαχείριση και ε, τη βάση δεδομένων των δικαιούχων για να δούμε πόσο εύκολο είναι να διαπιστώσουμε ποιες είναι οι φιλανδικές ΜΚΟ που παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πάρα πολύ ε, δύσκολη αυτή η δουλειά γιατί ε, στην Τράπεζα Δεδομένων δεν γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ των διαφόρων οργανώσεων. Αν κάνεις μια τέτοια έρευνα υπάρχει πληθώρα στοιχείων και ανακράτη μέλη, αλλά ποτέ δεν φαίνεται αν είναι ε, μη κυβερνητική οργάνωση συγκεκριμένη. Χρειάζεται και άλλη έρευνα. Κάναμε και αυτή την έρευνα, γιατί έχουμε πολλά στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τέσσερι διαφορετικέ υπηρεσίε. Europaid, ε, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον, το έχω για την ανθρωπιστική βοήθεια και Γενική Διεύθυνση Παιδεία και Πολιτισμού. Και φτιάξαμε τη δική μας βάση δεδομένων και μελετήσαμε πάρα πολύ προσεκτικά όλα αυτά τα στοιχεία για να είμαστε βέβαιοι ότι οι δικαιούχοι είναι μήκυο Και πού καταλήξαμε 1,4 δις ευρώ το 2009 περίπου. Είναι αύξηση των ε, αριθμών και των ποσών σε σχέση με το παρελθόν. Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλούσε για ένα δις περίπου για συνεργασία με ΜΚΟ. Και τώρα πρόκειται για τέσσερις και μόνο γενικές διευθύνσεις υπηρεσίες τις βασικότερες ως προς τον όγκο της συνεργασίας με ΜΚΟ. So you the βλέπουμε λοιπόν ότι το συνολικό ποσό, συνολικός όγκος ε, είναι στη Europe 8 κατά κύριο λόγο ε, μετά στο ε, έχω το Ευρωπαϊκό Γραφείο για την Ανθρωπιστική Βοήθεια και λιγότερο το περιβάλλον και η παιδεία και ο πολιτισμός. Τώρα, ως προς τον απόλυτο αριθμό των δωρεών, περίπου 3.000. 2.000 από τη Europaid και ακολουθούν η Έχω Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Παιδείας και Πολιτισμού. Δύο λόγια τώρα να σας πω για το γενικότερο πλαίσιο συνεργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ΜΚΟ το έτος 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ένα έγγραφο που περιέγραφε αυτή τη συνεργασία και τους βασικούς στόχους για τη συνεργασία αυτή. Και τότε η βασικότερη στόχη ήταν ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών γενικά και ε, ο τρόπος με τον οποίο ε, προβάλλεται αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλει εξέταση, πρέπει να ακούσουμε και ε, προσώπους κοινωνίας των πολιτών για να δούμε τι φρονούν εκείνοι και ε, ποια ήταν η συνεργασία ε, για την επιχειρησιακή της πτυχή όπου δεν μπορούν να είναι παρόντα τα κράτη ή ο ιδιωτικός τομέας έρχονται τα, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις και ε, υλοποιούν κάποια προγράμματα. Um, στη συνέχεια όμως δεν δόθηκε ακριβώς σωστή παρακολούθηση. Το 2000 έγινε πολύ εκτενής ε, και συνολική ε, παρουσίαση και αναφέρει και κάποια σημεία, κάποιες αδυναμίες ανατομέα, αλλά δεν δόθηκε συνέχεια. διαφέρει η συμπεριφορά και αντιμετώπιση των ΜΚΟ από γενική διεύθυνση σε γενική διεύθυνση και το προτείνουμε εμείς αυτό ε, ότι θα πρέπει να βελτιωθεί γιατί δεν έχουμε αρκετά στοιχεία που να ε, μαρτυρούν τι συνέχεια δόθηκε. Επίσης Ποιο είναι ο ορισμό των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι είναι δύσκολο να οριστούν διότι ε, διαφέρει το νομικό καθεστώ του καθενό ή τη κάθε οργάνωση σε κάθε κράτο μέλο. Ε, και θα πρέπει να ε, δούμε με ποιο τρόπο οι Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπηρεσίε διαχειρίζονται καν αυτέ τι εταιρείε. Ούτε εκεί είναι ενιαία η διαχείριση και η αντιμετώπιση ποιο θεωρεί μη ποιον. Ο βασικός χαρακτήρας είναι η μη κερδοσκοπική βεβαίως διάσταση, αλλά και κάποια άλλα στοιχεία. Να υπάρχει ένα νομικό καθεστώς, ε, να υπάρχει ένα είδος εθελοντισμού, έτσι, εθελοντικής εργασίας και να είναι ανεξάρτητη βεβαίως από κυβερνήσεις η οργάνωση αυτή. Α, μήπως να δώσω τώρα το λόγο στον συνάδελφό μου να μας πει κάτι για την αποτελεσματικότητα και την ε, αποδοτικότητα αυτών των ε, μέτρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε που μας δίνει δυνατότητα να σας κάνω αυτή την παρουσίαση. Ήταν ενδιαφέρον στην αρχή να δούμε ποιο είναι το λεξιλόγιο που χρησιμοποιήθηκε, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα χρησιμοποιήθηκε. Αυτή η όρη είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τον έλεγχο. Περί αυτού πρόκειται. Όταν μιλήσαμε με τις ΜΚΟ, προσπαθώντας να πάρουμε απαντήσεις σχετικά με την εμπειρία τους από τη συνεργασία τους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις συμβάσεις για τις χωριές, τότε αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε τι μπορούν να κάνουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση οι ΜΚΟ. Πώς μπορούν να βοηθήσουν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό πλαισιώνεται από τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται. Μας ανέφεραν κάποια προβλήματα. Τις διάφορες λεπτομέρειες, τις τυπικές ανέφεραν. Το είπε και ο Σιτάλα. η χρονική περίοδος κατά την οποία παρέχει υποστήριξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η χρηματοδότηση που βασίζεται στα προγράμματα είναι η βασική προσέγγιση που ακολουθείται και σύναψη συμβάσεων. Και τα πλέον μακροπρόθεσμα προγράμματα και χρηματοδότησή τους. Δεν σημαίνει ότι αένα χρηματοδοτούνται τα προγράμματα, πιστεύουν ότι η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση τις βοηθάει καλύτερα να πετύχουν κάποιους στόχους που τις απασχολούν. Μπορούν να εστερνιστούν τα προγράμματα που εφαρμόζουν έτσι έναντι των δικαιούχων. Και αυτό σχετίζεται με το σωστικό στόχο, την αποτελεσματικότητα. Ποιο πρόβλημα θέλει να λύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να διαλέγει ΜΚΟ που μπορεί να τη βοηθήσουν. Είναι παροχή υπηρεσιών ο τελικός στόχος και η βελτίωση όσον αφορά τα δικαιώματα διαφόρων κοινοτήτων και ατόμων. Άρα θέλουμε αποτελεσματικό όσον αφορά τους μακροπρόθεσμους στόχους. Εκεί χρειάζεται βελτίωση, είπαν οι ΜΚΟ, μέσω μακροπρόθεσμων διευθετήσεων χρηματοδοτήσεως και χρηματοδοτήσεως προγραμμάτων άλλη πτυχή που έφυξαν. Τις δυνατότητες που έχουν οι φορείς αυτοί, οι ΜΚΟ, για να κάνουν τη δουλειά τους. και που αλλάζουν οι περιστάσεις μετά από μια χρονική περίοδο. Άρα πολύ βραχυπρόθεσμο πλαίσιο χρηματοδοτήσεως με πολύ μεγάλους περιορισμούς όσον αφορά τους στόχους και τα αποτελέσματα ίσως δεν τους παρέχει την αναγκαία ευελιξία για να μπορέσουν να πετύχουν τους ευκταίους στόχους. Χρειάζεται ισορροπία. Το αναγνωρίζουν οι ΜΚΟ. Και εκεί θέματα που προαναφέρθηκαν και αναφέρονται και στο έγγραφο. Πώς προωθείται η καινοτομία. Πώς αποφεύγεται φυσικασμός. Πώς αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα. Και πώς βρίσκονται νέες λύσεις. μας ανέφεραν διάφορα στοιχεία η ΜΚΟ. Όχι μόνο η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων, αλλά και ο μηχανισμός επιλογής αναφέρθηκε. Οι γενικές διευθύνσεις έχουν τον πρώτο λόγο όσον αφορά τις προσεγγίσεις που ακολουθούνται. Ίσως χρειάζεται εναρμόνιση μεταξύ των γενικών διευθύνσεων. Έτσι θα είναι πιο εύκολη η πρόσβαση των ΜΚΟ στα συστήματα. Αναφέρθηκα στην περιορισμένη ευελιξία που θεώρησαν οι ΜΚΟ ότι υπάρχει και ότι θέλαν περισσότερο χώρο να κινηθούν. Και κάτι σημαντικό. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά τους φορείς αποδέκτες. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι ανάλογοι των μεγεθών των ΜΚΟ. Οι μικρές ΜΚΟ που αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα για να μπορέσουν να προωθήσουν καινοτόμα στοιχεία στη σχέση που έχουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος. Μία επισκόπηση των πορισμάτων όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Πώς παρουσιάζονται, πώς υπάρχει ενημέρωση για αυτά. Βλέπετε ένα πίνακα. Ο πρωταρχικό τρόπο ενημέρωση και αξιολόγηση και υποβολή εκθέσεων όσον αφορά την αποτελεσματικότητα τη λειτουργία των φορέων αυτών που χρηματοδοτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η αυτοαξιολόγηση. Αυτό συνεπάγεται διάφορα ωφέλη για τους φορείς αυτούς, αλλά και μειονεκτήματα. Θα πρέπει να γίνεται κάποια εξακρίβωση των διαφόρων ισχυρισμών που γίνονται στα πλαίσια της αυταξιολόγησης. Όπως είπε και ο Σμπρουμάια προηγουμένως, η μελέτη μας βοήθησε να δούμε που υπάρχει καλή πρακτική όσον αφορά την χρήση εξωτερικής αξιολογήσεως από τρίτα, τρίτους φορείς όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν ένα παράδειγμα της Ολλανδίας ακόμα και όταν κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έχουν διάφορες πρακτικές που εφαρμόζουν, που ξεπερνούν την αρχή της αυτοαξιολογήσεως. Ήταν ένα παράδειγμα αυτό. Αυτό βοηθά, σαν παράδειγμα. Να χρησιμοποιούμε επικύλα εργαλεία για την αξιολόγηση. Πριν ξαναπάρει το λόγο και ο Μπρουμάιερ, θέλω να πω κάτι. Είδαμε και διαπιστώσαμε ότι τα εργαλεία που υπάρχουν και το σύστημα διαλόγου και επαφής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τους αποδέχτες των χωριών λειτουργεί εν γέννη. Γενικό αίσθημα που επικρατεί είναι ότι οι ουσιαστικοί στόχοι επιτυγχάνονται, οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και διευκολύνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευρύνει την εισρωή πληροφοριών η διαμόρφωση πολιτικής. Και αυτή είναι από τις βασικές συμμετοχέ της κοινωνία των πολιτών. Τέλος. Κάτι επανέφερε ο κ. Μπρούμαγερ. Οι οργανώσει κοινωνία των πολιτών και ΜΚΟ είναι φορεί που ξεπερνούν κατά πολύ τη σφαίρα επιρροή των κυβερνητικών και δικυβερνητικών δομών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Γενικά η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική. Σε άλλους τομείς χρειάζεται να γίνουν πολλά και διάφορα πράγματα και ελπίζω ότι καταφέραμε να ξεθάψουμε πολλά από αυτά που πρέπει να γίνουν. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ ζήτησε το λόγο. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Δεν τελειώσαμε ακόμα, δεν τελειώσαμε. Πέντε λεπτά να μου δώσετε. Και μετά η κυρία Γιάλα Σέντερ θα πάρει το λόγο. Λίγα πράγματα για το θέμα της διαφάνειας συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωση και ΜΚΟ. Το είπα και πιο πριν και το είπε και ο κύριος Ήταλα. Το σύστημα οικονομικής διαφάνειας δεν, δεν δίνει τη δυνατότητα να καταγράφονται οι ΜΚΟ. Απλώς μπορεί να πει ότι ε, αυτό το κράτος μέλος, ε, αυτή η Φιλανδία, πήρε αυτή την χρηματοδότηση αλλά δεν μπορεί να δει ποιος είναι ποιες είναι, ποιοι είναι οι δικαιούχοι ουσιαστικά. Δεν υπάρχει διαχωρισμός, ανατύπω χορηγίες, δεν φαίνεται για ποιο λόγο έχουν χρησιμοποιηθεί τα κονδύλια αυτά. Και επίσης δεν υπάρχει και απόλυτη ορατότητα αυτών των δεδομένων. Σε όλες τις γενικές διευθύνσεις βεβαίως μπορούμε να βρούμε στο τέλος της τις ε, πληροφορίες, ε, είμαστε γνώστες του πώς βλέπει το σύστημα της Κομισιόν, αλλά για έναν που δεν έχει εμπειρία δεν θα είναι τόσο εύκολο. Ίσως να είναι πιο εύκολο να υπάρχει ένα, μια ενιαία θηρίδα, ένα ενιαίο σημείο εισόδου. Και βλέπετε εδώ στη διαφάνεια ότι όλες οι υπηρεσίες που είδαμε λεπτομερέστερα ε, δημοσιεύουν τις πληροφορίες για τις μη που, που επωφελούνται των χρηματοδοτήσεων. Ε, τρεις περιπτώσεις μόνο υπήρχαν διαφορετικές, που ήταν για μη κερδοσκοπικές ε, κυβερνητικές οργανώσεις. Τώρα για την εκπροσώπηση ε, και για το πώς χρησιμοποιούν το σύστημα η καπαόμικρον. Είδαμε ότι το χρησιμοποιούν σωστά. Αποτελούν περίπου το 39% των, ε, των εισόδων από τον ε, Σεπτέμβρη το ποσοστό, όπως βλέπετε, έχει ε, αυξηθεί. Βλέπετε ένα κράτος μέλος και ποιες είναι οι ΜΚΟ. Κυρίως βλέπετε από το Βέλγιο πολλές. Υπάρχουν και ευρωπαϊκά δίκτυα ΜΚΟ που είναι εδώ πέρα στις Βρυξέλλες, οπότε είναι λογικό. Αλλά είδαμε ότι οι ΜΚΟ και κυρίως αυτές που δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητες ε, lobbying στην ε, ε, Κομισιόν. Από τις 120 που απαντήσανε στην έρευνα, είδαμε ότι μόνο ένα, ένας μικρός αριθμός είπε ότι ναι, εμείς κάνουμε lobbying, αλλά δεν έχουμε καταχωρηθεί. Είναι κάποιες, αλλά είναι πολύ μικρό το μερίδιο της πίτας που τους αναλογεί. και δεν ε, έχουν πάρει μέρο σε καμία δραστηριότητα διαφάνειας. Για τα συμπεράσματα τώρα. Καλό θα ήταν να ενημερώσουμε το πλαίσιο που υπάρχει από το 2000 που έχει η Κομισιόν για να δούμε πώς μπορούμε να μελετήσουμε δυνατότητες δημιουργίας μιας ε, συγκεκριμένης ε, ομοιογενούς ορολογίας, τι μπορούμε να κάνουμε για να εναρμονίσουμε το σχεδιασμό το, και την λειτουργία της ε, όλης διαδικασίας χρηματοδότησης ε, των ΜΚΟ. Είχαμε και την, ε, και την μελέτη που έγινε ανά υπηρεσία και ίσως να πρέπει να τεθούν και κάποια όρια στη χρηματοδότηση. Αν δείτε ποιο είναι ο στόχο τη ε, Κομισιόν, να διευρύνει τι πολιτικέ τη, να συμπεριλάβει τι ε, ΜΚΟ στην ε, διαδικασία, αλλά από ό,τι φαίνεται οι ΜΚΟ είναι εξαρτημένε και μάλιστα πολλέ ασκούν και κριτική, γιατί εξαρτώνται πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και μπορεί, αυτό, μπορεί κάποιο αυτό να αμφισβητήσει την ανεξαρτησία του, εφόσον εξαρτώνται τόσο πολύ από την Κομισιόν. Και αυτοί που το κατάλαβαν αυτό είπαν ότι θα πρέπει ίσως να περιορίσουμε τη χρηματοδότηση. Ή θα πρέπει, αν, μπούμε σε, αν εξασκούμε δραστηριότητες ε, lobbying, να μην λαμβάνουμε ε, χρηματοδότηση από την Κομισιόν. Να επαναλάβω τις συστάσεις που προέκυψαν από την ε, μελέτη μας. Αυτό λοιπόν που προτείνουμε είναι να... Εντάξει, βελτιώθηκε βέβαια η χρήση του προγράμματος χρηματοδότησης, αλλά να διευρύνουμε το πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα να τεθεί σε ένα, σε ένα πλαίσιο αυστηρών διαδικασιών εφαρμογής, ελέγχου και αξιολόγησης μεταξύ, μέσα στα πλαίσια ενός διαλόγου μη καπαόμικρων και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ βλέπετε ε, το ενδιαφέρον που υπήρξε για μια τέτοια πιο στενή συνεργασία. Τώρα, στη φορά την επάρκεια, εμ, υπάρχει προστιθέμενη αξία μέσω μιας πιο συστηματικής ε, ε, αξιολόγηση συγγνώμη, της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας με τις ΜΚΟ, μπορούμε να στοχοθετήσουμε τις εφαρμογές, την, ε, τον έλεγχο και όλες τις σχετικές διαδικασίες μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων και επίσης μπορούμε να θέσουμε συγκεκριμένες απαιτήσει για την υποβολή εκθέσεων και τον έλεγχο που θα μπορούν να γίνουν έτσι λίγο πιο αναλογικές ανάλογα με το μέγεθος του, της χορηγίας, της δωρεάς. Και Τέλος. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, προτείνουμε να μειωθεί η, αυτή η μεγάλη εξάρτηση από την αυτοαξιολόγηση και να ενισχύσουμε την εξωτερική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συνεργασίας ε, ε, ε, ε, ε και ΜΚΟ. Για τα θέματα διαφάνειας, καλό θα ήταν να εναρμονίσουμε την παρουσίαση των, ε, των πληροφοριών που έχουμε για την χρηματοδότηση, γιατί τώρα γίνεται με τελείως καταγερματισμένο τρόπο αυτό, γιατί υπάρχουν οι πληροφορίες, αλλά η χρησιμότητά τους ίσως είναι περιορισμένη τώρα. Θα μπορούσαμε ίσως να δίνουμε πληροφορίες ανάλογα με τον τομέα, με την γενική διεύθυνση κτλ. Και επίσης θα μπορούσαμε να δούμε κατά πόσο το ε, μητρό των ε, ενδιαφερομένων εκπροσώπων θα μπορούσε να ενισχυθεί. Αυτοί δηλαδή που δεν έχουν καταγραφεί, καταχωρηθεί, να το πράξουν. Να δούμε ποιες είναι οι κατηγορίες ε, οργανώσεων που θα πρέπει να καταχωρηθούν. Και σε ό,τι αφορά τον ποιοτικό έλεγχο, το είπαμε και πιο πριν αν δείτε την ε, βάση δεδομένων, συχνά υπάρχουν έτσι κάποια απλά λάθη. Ας πούμε κάποιος γράφει μια λάθος χώρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό λίγο μειώνει και την ε, επαγγελματική άποψη που θα έπρεπε να δείχνει αυτός, αυτό το μητρό. Να αυξήσουμε την ε, ορατότητα του RIR μέσω των, ε, οργανώσεων, των γενικών οργανώσεων ΜΚΑ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την παρουσίαση. Πριν δώσω το λόγο συναδέλφους, θα ζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν θέλει να παρέμβει. Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τη Γενική Διεύθυνση Υπολογισμού είμαι. Ευχαριστώ στον συγγετή και στου εμπειρογνώμονε που έκανα την πολύ λεπτομερή παρουσίαση τη μελέτη. Την περασμένη εβδομάδα λάβαμε γνώση αυτή. Έχετε μπροστά σα μια αντιπροσωπή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει εκπρόσωπο τη Γενική Γραμματεία, κ. Γκρι, τη Γενική Διευθύνσεω ΚΟΜ, την κυρία Λεκλέρκ, τη Γενική Διευθύνσεω Περιβάλλοντο, τη Γενική Διευθύνσεω ΔΕΦΚΟ και τη Γενική Διευθύνσεω ΕΚΟ. Όλε οι γενικέ διευθύνσει ακούστηκαν, αν θέλετε, εξέφρασαν απόψεις για τη διαμόρφωση της μελέτης και οι συνάδελφοι θα θέλουν, πιστεύω, να προβούν σε κάποιες ευκρινήσεις και να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις σας. Ε, εν συντομία, σημειώνουμε, κύριε Πρόεδρε, την ύπαρξη της μελέτης αυτή. Συμφωνούμε επί του γενικού τόνου που ακολουθείτε και επί των τάσεων που ακολουθούν οι συστάσεις και οι παρατηρήσεις της εκθέσεως. Σημειώσαμε όμως και κάποια θετικά σχόλια και περιθώριο για βελτιώσεις. Υπάρχουν και κάποια θέματα που αναφέρονται επανειλημμένα, αλλά είναι εξίσου σημαντικά. Το θέμα της διαφάνειας, το θέμα της ελήψεως ή όχι ορισμού για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση, όλες αυτές οι συστάσεις σωστά αναφέρονται εδώ, γιατί ξεκινούν οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής την προετοιμασία της νέας γενιάς των προγραμμάτων και λαμβάνουμε υπόψη ως τις παρατηρήσεις στα πλαίσια των εργασιών αυτών. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Θα συζητήσουμε αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο που το FTS, το Financial Transparency System, σύστημα οικονομικής διαφάνειας που υπάρχει από το 2008 και ζήτησα από τους αρμόδιους συναδέλφους να μιλήσουν. Είναι αρκετά δημοφιλές περίπου 20.000 με 60.000 hits στο διαδίκτυο, χτυπήματα στο διαδίκτυο το μήνα. Αναφέρθηκε ότι μέχρι τώρα δεν υπήρχε δυνατότητα να εντοπίζονται οι δικαιούχοι κατά κατηγορία. Είναι κάτι που το συζητήσαμε στα πλαίσια της απαλλαγής του 2008. Το Κοινοβούλιο μας έκανε συστάσεις σχετικές. Θα τις ακολουθήσουμε. Επεξεργαζόμαστε αυτό το εργαλείο λοιπόν και παίρνουμε τα στοιχεία και μέχρι το 2011 θα έχουμε ένα πεδίο non-profit organizations και profit organizations, Μη κερδοσκοπικού και κερδοσκοπικού οργανισμού και φορεί. Μέχρι το 2013 θα υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό στα πλαίσια του εργαλείου FTS, λοιπόν. Ευχαριστώ. Η συνάδελφο Αγιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τη μελέτη αυτή. Πολύ εμπεριστατωμένη για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες μας ε, για τη στιγμή που καλούμαστε να αποφασίσουμε το πώς ε, θα ελέγχουμε τη χρηματοδότηση το ΜΚΟ και κυρίως πώς θα αυξήσουμε και την επάρκειά τους και την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητά τους. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις των μελετών βλέπω ότι επικεντρώνονται κυρίως, τουλάχιστον από αυτά που μπόρεσα εγώ να καταλάβω, γιατρώνονται, λέω στην Ισπανία και την Ολλανδία. Και θα ήθελα να ρωτήσω γιατί υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος που ε, επιλέξατε ακριβώς αυτά τα δύο κράτη. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα κράτη που δίνουν το 50% της ενίσχυσης της ΜΚΟ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια Γιατί επιλέξατε αυτές τις δύο χώρες και γιατί αφήσατε απ' έξω άλλες οργανώσεις που συχνά ε, μας απασχολεί εάν χρηματοδοτούν ε, τα ε, προγράμματα αυτά για καλό ή για κακό γιατί είναι ένα λόμπι στη συνέχεια που αντί να μας διευκολύνει μας δυσκολεύει τη δουλειά μας και μετά γιατί τη χρηματοδότηση. Ιστορικά εδώ έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα στην Επιτροπή μας στη συγχρηματοδότηση ε, διεθνών ε, οργανισμών. Είτε πρόκειται για την Παγκόσμια Τράπεζα, για τα Ηνωμένα Έθνη και πάντα προσκρίουμε σε κάποια διαφάνεια και κρυψίνια όταν ε, θέλουμε να ελέγξουμε τα προγράμματα. Πάντα είχαμε προβλήματα και προσκόμματα στην άλλη πλευρά στη συγχρηματοδότηση επαναλαμβάνω για τη Ολλανδική διοίκηση φέρεται ως θετικό ε, σημείο τη δυνατότητα να γίνει αλλαγή στα προγράμματα των ΜΚΟ, δηλαδή επέμβαση του χρηματοδότη. Ξέρετε ότι τώρα γίνεται μια μεγάλη συζήτηση. Αν θα πρέπει να πάμε προς ένα μοντέλο συγκέντρωσης των ΜΚΟ σε συγκεκριμένους ε, τομείς, και εδώ υπάρχει κίνδυνος να μην βοηθούμε επιτόπου της ΜΚΟ που χρειάζεται και κάποια αποκέντρωση ή κάποια διασπορά. Ή το αντίθετο, να παραμένουμε σε αποκεντρωμένη διαχείριση, πράγμα όμως που δυσκολεύει τη χρηματοδότηση, έχουμε επικαλύψεις, επαναλήψεις και προβλήματα. Για να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε όλα αυτά χωρίς να έχουμε τεράστια προβλήματα και κινδύνους να χάνουμε την αποτελεσματικότητά μας. Ευχαριστώ. Κύριος Χατζημαρκάκης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με εκπλήσει πάρα πολύ που δεν έχουμε ακόμα ορισμό το τι είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Στην ακρόαση θα θυμούνται κάποιοι συνάδελφοι που κάναμε με τον Επίτροπο Σεύσκοβιτς, είχαμε προειδοποιήσει και από ό,τι φαίνεται ακόμα δεν έχει προκύψει ε, ενιαία αντίληψη, δόγμα, όραμα, τι στη ΜΚΟ. Για μένα είναι πρόβλημα αυτό. Άμα δεν ξέρω ποιος είναι αυτός, πώς να συναλλαγώ μαζί του. Ε, έχουμε πληθώρα διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων με πληθώρα διαφόρων ε, υποθέσεων που είναι πολύ σημαντικές αλλά κάποιες άλλες είναι τελείως ασήμαντες. Υπάρχει ΜΚΟ ας πούμε που ε, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μόνο που κάνει είναι να λιδωρεί και να κατηγορεί συνέχεια ε, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει εμείς να υποστηρίζουμε οικονομικά ε, αμερικανικής ε, κοπής ΜΚΟ που μας υπονομεύουν και μας κατηγορούν. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Είναι εκπρόσωποι συμφερόντων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να καταλήξουμε τι εστί μη κυβερνητική οργάνωση. Κάτι άλλο που με ενοχλεί επίσης λίγο και ευχαριστώ τους κυρίους για τη μελέτη που μας παρουσιάζουν είναι ότι δεν υπάρχει ενιαία επισκόπηση. Εντάξει, μιλήσατε για μια δημοσίευση του 2008, αλλά θα πρέπει κανείς να βρει το δρόμο του στις διάφορες ε, γενικές διευθύνσεις και χρειάστηκε πάρα πολύ χρόνο και για μας τους βουλευτές να πάρουμε απάντηση από τις γενικές διευθύνσεις για το ποιους... Εμ, υποστηρίζουν και ποιου ε, χρηματοδοτούν. Γιατί μα παραπέμπουν στι γενικέ διευθύνσει. Πηγαίνετε και ρωτήστε τι υπηρεσίε αυτοί του χρηματοδοτούν, αυτό το διαχειρίζονται. Ε, δεν πάει έτσι όμω, γιατί είπαμε θα πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η επάρκεια του, ποια είναι η λειτουργία του, ποια είναι η αποτελεσματικότητά του και θέλουμε να έχουμε μια ενιαία εικόνα. Επίση, κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω. Μια κατάσταση. Ακριβώ επειδή είναι τόσο κατανεμημένα αυτά στι γενικέ διευθύνσει, που καταρχήν δεν έχω πρόβλημα αλλά να κάνω μια παρένθεση, να έχουμε μια ενιαία έτσι, τυποποιημένη θεώρηση για τις ΜΚΟ, κλείνει παρένθεση. Έχω την εντύπωση ότι παίζει ο ένας επίτροπος ενάντια στον άλλον και η Γενική Διεύθυνση το διαπίστωσε αυτό στο περιβάλλον. Έχουμε επιτρόπους ε, που συνδέονται με το περιβάλλον και είναι επίτροπος για την προστασία του κλίματος ή επίτροπος για ε, το περιβάλλον βασίζονται και επικαλούνται μελέτες ΜΚΟ για να στραφούν κατά του έργου άλλων επιτρόπων. Βλέπετε τη βιομηχανία. Ε, εντάξει, και αυτό καλό, αλλά είναι αποτελεσματικό. Αυτό μας βοηθάει στη δουλειά μας. Θεμητό μπορεί να είναι, αλλά δεν θα μπορούσαμε καλύτερα να ε, ε χρησιμοποιούμε τα κοινοτικά κονδύλια και τις πιστώσεις. Χαίρομαι για τη μελέτη αυτή, πραγματικά ήταν χρόνος να γίνει αλλά παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει και τις συστάσεις και τις προτάσεις και να τα λάβει σοβαρά υπόψη της. Ο Επίτροπο Σεύσοβιτ, νομίζω, ω αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα λαμβάνει όλα αυτά πολύ σοβαρά υπόψη. Τουλάχιστον αυτό απορρέει από τι συνομιλίε που είχαμε και την περασμένη εβδομάδα που είχε έρθει στην Επιτροπή μα για άλλο θέμα. Παρ' όλα αυτά έρχεται τακτικά και τα συζητάμε. Και εναπόκειται και παραμένει το αίτημά μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, γιατί αλλιώ δεν μπορούμε να εξηγούμε στους φορολογούμενους τι χρηματοδοτούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριος Γκέιρ, έχει το λόγο. Σύντομα, Πρόεδρε. Έθεσαν πολλά ερωτήματα οι συνάδελφοι. Ένα σχόλιο και μια ερώτηση από μένα. Αυτό αυτή την αυτοαξιολόγηση δεν την καταλαβαίνω εγώ ιδιαίτερως, με προβληματίζει. Γιατί νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα πώς κάποιος από την που λαμβάνει χρήματα από την Κομισιόν μπορεί να, εντάξει, μπορεί με να αξιολογηθεί εξωτερικά, αλλά τουλάχιστον εγώ έτσι κατάλαβα, σε ό,τι αφορά την ε, αυτοαξιολόγηση, αυτή η αξιολόγηση πρέπει να πει πόσο αποτελεσματικά έχει χρησιμοποιήσει τα κονδύλια. Αυτό πώς, πώς μπορεί κάποιος να είναι τόσο αντικειμενικός. Εγώ δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά ή λάθος. Αν κατάλαβα λάθος με διορθώνετε. Ευχαριστώ, έχει το λόγο για τι απαντήσει. Θα πάω στο τελευταίο ερώτημα. Είναι θέμα παρουσιάσεω ε, PowerPoint, μετατροπής των αρχείων από PowerPoint σε Mac. Η κυρία Αγιάλα ρώτησε γιατί επιλέξαμε την Αγενσία Σπανιόλα Κοπερασιών. Το συζητήσαμε αυτό με τους αρμοδιούς που μας, μας το ζήτησαν αυτό, βάλαμε στην έκθεση παραδείγματα από άλλα κράτη-μέλη. Όπως ανέφερα, ήρθε μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και αυτό μας περιόρισε και οι πόροι μας ήταν περιορισμένοι. Έπρεπε να εξετάσουμε μόνο δύο κράτη-μέλη. Επιλέξαμε την Ολλανδία, διότι ακολουθούσαν καινοτόμε ε, προσεγγίσεις όσον αφορά τι ΜΚΟ και επέλεξα την Ισπανία γιατί ζω στην Ισπανία, μένω στην Ισπανία. Μέχρι εκεί φτάσαμε. Δεν μπορούσαμε να διευρύνουμε το πλαίσιο Θέλαμε να συλλέξουμε κάποιες βέλτιστες πρακτικές. Ίσως να αποτελούσαν έμπνευση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν συμπεριλαμβάναμε αυτές τις πρακτικές στην έκθεση, στη μελέτη. Ίσως δεν διαρευνήσαμε κάποια ζητήματα πλήρως ότι χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα, κάποιες ΜΚΟ και να αντιπαρατίθεται κάποιες ΜΚΟ μεταξύ τους. Δεν το εξετάσαμε λεπτομερώς. Υπήρχαν κάποια προβλήματα. Είδαμε άρθρα, ερωτήσεις. Γιατί να δίνουμε χρήματα σε μία ΜΚΟ που έρχεται σε κάποια σημαντική συνάντηση και μας επικρίνει. Αυτό δεν είναι μόνο τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στην Παγκόσμια Τράπεζα και σε κάποια κράτη-μέλη έχουν παρόμοια θέση. Υπάρχει αυτό συμβαίνει. Θέλουμε οι ΜΚΟ να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για να εξισορροπήσουν τις απόψεις που εκφράζονται με ισχυρότερο τρόπο από τη βιομηχανία, από πιο ισχυρούς εμπλεκόμενους. Άρα γίνεται δεκτό αυτό. Ο Μάικλ, Μάικλ θες να πεις κάποια πράγματα για τα άλλα ζητήματα, την ευελιξία κλπ. Ναι. δεν ασχοληθήκαμε εις βάθος και ειδικά με τη σχηματοδότηση. Αλλά ανέκυψε. Ναι, Όταν έχουν προσφορά χρηματοδοτήσεως οι οργανώσεις είναι ένα πρόβλημα, κυρίως στην ισχύουσα οικονομική κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουν τα πρώτα χρήματα που χρειάζονται για να φτάσουν στη δεύτερη δόση. Μέσω του μηχανισμού αποκλείονται τελικά από τη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πετύχουν κάτι που θέλουν και οι δύο πλευρές. Πρέπει να εξεταστεί ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να επιτευχθεί ένας κοινός στόχος. Σωστά τίθεται τα ερωτήματα για την χρήση της χρηματοδοτήσεως, κυρίως όταν αφορά πολύ μεγάλα ποσά. Τώρα, οι διάφοροι ορισμοί του τι αποτελεί μη κυβερνητική οργάνωση. Είναι ένα μη ορισμό. Είναι μη κυβερνητική οργάνωση. Ο φυστάμενο ορισμό είναι τι δεν είναι. Αυτό λέει πολλά για το πώς υπάρχουν αντιφάσεις όσον αφορά το ρόλο τους και τις σχέσεις τις χρηματοδοτικές που υπάρχουν. Υπάρχουν φορείς που παρέχουν μια υπηρεσία για διάφορες πολιτικές αλλά ίσως να μην εξυπηρετούν πάντα στατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό θα το απαντήσουμε εμεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα σταθμίσουν αυτά. Το θέμα των μικρών μη κυβερνητικών οργανώσεων και πώ έχουν πρόσβαση. Και το θέμα του κόστους των συναλλαγών. Είναι θέμα επίτευξης πολιτικών στόχων. Ίσως θα θέλουν να το εξετάσουν αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. ένα από τα πιο γενικά ζητήματα που αφορούν τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ είναι ότι όλο και περισσότερο επιτρέπουν στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαμόρφωση πολιτικών που τους επηρεάζουν. Αυτό είναι γενικά θετικό. Και κάθε βουλευτής είναι δίωδος αν θέλετε που, από την οποία περνούν τα συμφέροντα των πολιτών. Και αν συμφωνούν με αυτό θέλουν αυτός ο διάβλος παραμείνει, αυτή η διάβλος να παραμείνει ανοιχτή. Σκέψη είναι και όχι σύσταση. Η απάντηση είναι πολύ δύσκολο να δοθεί, γενική απάντηση. Κάθε χώρα ίσως χρειάζεται διαφορετική απάντηση, ανάλογα με τη φάση εκδημοκρατισμού στην οποία βρίσκεται και ανάλογα με σας παράγοντες που ισχύουν. Ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις.